Καλησπέρα σας. Ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας. Το πρώτο σημείο είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης και εάν δεν υπάρχουν αλλαγές, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Δεύτερο σημείο, ανακοινώσει Προέδρου. 2-1. Συστάσει στι οποίε προβαίνουν οι συντονιστέ. Μετά από τη συνεδρίαση τη 20 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια δια τη γραπτή διαδικασία στις 7 Μαρτίου οι συντονιστές αποφάσισαν να συντάξουν μία προφορική ερώτηση με, ψήφισμα για τον προϋπολογισμό και το φύλλο και να το χορηγήσουν στην ομάδα ALDE, να συντάξουν νομοθετική γνωμοδότηση ε, υπό τον κανονισμό κανόνα 53 για την πρόταση κανονισμού για την αξιολόγηση ε, της τεχνολογίας ε, ε βοηθές και να διζητήσουν διοδότηση για ε, έξι αποστολές και πέντε ακροάσεις για το δεύτερο ήμιση του 2018. Επόμενο σημείο, να σας καλωσορίσω τα νέα μέλη της Επιτροπής μας και να καλωσορίσω τον κύριο Ζερόμα ε, Λαύρη από την ομάδα του ΕΛΚΑ που ήρθε στην Επιτροπή μας ως αντικαταστάτης, ως πληρωματικό μέλος, σε χαρτίρια και σας ευχόμαστε να συνεργαστούμε πολύ ε, καλά εδώ στην Επιτροπή μας. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων για το Δεκέμβριο 2017, 4 Δεκέμβριο 2017, αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνονται τα πρακτικά. Επόμενο σημείο, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, αγαπητοί συνάδελφοι, είστε έτοιμοι. Έχετε τις ε, κάρτες σας για τις ψηφοφορίες. Σημείο 4 της ημέρης διάταξης. Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης. Ε, πρόκειται για την έγκριση του σχεδίου θέσης υπό τη μορφή τροπολογιών. Η συγγήτρια είναι η κυρία Αγγέλικα Μλίναρ. Και θα ξεκινήσουμε τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, ε, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 με προφορική τροπολογία την οποία ζήτησε το ΕΛΚ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στην κυρία Συγγνώμη, διακόπτει η, η Πρόεδρος. Ναι, βεβαίως να αλλάξουμε την 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ την κυρία Μλίναρ. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ψηφοφορία επί του εξυγχρονισμού της εκπαίδευσης στην Ένωση. Η ε, υιοθέτηση του σχεδίου γνωμοδότησης της κυρίας Σοντρόβα. συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 σε τμήματα. Α, μόνο το δεύτερο τμήμα. Ναι. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45, τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θέλετε να ελέγξουμε την 54 Ωραία. Να ελέγξουμε την 54. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά παρακαλώ να ελέγξουμε. 56. Άρχεται η ψηφοφορία. Και τώρα τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ να ελέγξουμε. 55. Ε, άρχεται η ψηφοφορία και τώρα Τελειώνει. Ε, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά άρχεται τέλος εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 73. And now the Τέλος. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος, μάλιστα. 74 ελέγχουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Γιατί 12 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. 12. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 16. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ αποχές ε, κατά αποχές ε, εγκρίνεται 25 υπέρ κατά Αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την τοπολογία 25. Τέλος πληροφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σχέδιο της νομοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στην εισηγήτρια Μιχαέλα Σοντρόβα. Δεν έχουμε άλλες ψηφοφορίες στην ημερήσια διάταξη και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 Συνάδελφοι, ας περάσουμε στο σημείο 6, η αποστολή στην Ουγγαρία. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται η έκθεση αυτή. Και στις 3 υποδεχθούμε την Επίτροπο Γιούροβα, υπεύθυνη για ζητήματα δικαιοσύνης καταναλωτών και ισότητας ε, των φύλων. Ε, θα γίνει μια ανταλλαγή απόψε με την Επίτροπο για στα πλαίσια του διαφορετικού διαλόγου, διαθρωμένου διαλόγου. Θα περιμένουμε λοιπόν μερικά λεπτά μέχρι να φτάσει η Επίτροπο. Συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε τώρα την ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο του διαφθορμένου διαλόγου με την Επίτροπο Βέρα Γιούροβα. Όπως ε, κάθε χρόνο η Επίτροπος ε, επισκέπτεται την Επιτροπή μας στο πλαίσιο του διαφθορμένου διαλόγου και έχουμε Έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λοιπόν με την Επίτροπο τα βασικά ζητήματα που άπτονται των δικαιωμάτων των γυναικών και υπάγονται στο δικό της χαρτοφυλάκιο. Το νέο σχέδιο δράσης ε, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ άντρων και γυναικών θα είναι ένα από τα κύρια ζητήματα σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων, καθώς και ε, οι δέσμοι μέτρων για την ε, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού βίου. Τα δύο αυτά θέματα, καθώς και η εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και στο πλαίσιο φυσικά της πρόσβασης Ευρωπαϊκής, ε- προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και η προώθηση ε, των γυναικών σε ε, ρόλους και σε θέσεις ευθύνης είναι προτεραιότητες για μας. Δίνουμε λοιπόν το λόγο στην Επίτροπο. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Μόλις σε μερικές εβδομάδες πέρασαν από την τελευταία μας ε, συνάντηση ε, κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας και είπα ότι θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο και ενέργεια στα ζητήματα της ισότητας ε, μεταξύ των φίλων για πάνω από μία μέρα το χρόνο. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε αυτή τη δυνατότητα σήμερα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα σήμερα να σταθώ ε, στις βασικές εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ισότητας των φύλων. Πρώτον, κλείνοντας ε, το έτος 2017 με σχεδιασμένες δράσεις για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, ε, ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για την εξάλληψη αυτού του φαινομένου. Δεύτερον, έχουμε το σχέδιο δράσης για, για την ισορροπία μεταξύ προσωπικού και επαγγελματικού βίου, το συνέδριο του 2017 για τα θεμελιώδη δικαιώματα που ε, ασχολήθηκε ακριβώ με την ισότητα των φύλων και η πρώτη σύνοδος κορυφής G7 ε, με βασικό θέμα την ισότητα των φύλων, στην οποία συμμετείχα εκπροσωπώντα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, όπως ανακοίνωσα εδώ την περασμένη φορά, Υιοθετήσαμε το σχέδιο δράσης 17-19 για να καταπολεμήσουμε το μισθολογικό χάσμα. Θα ήθελα τώρα να επισέλθω σε ό,τι αφορά αυτό. Το 2017 ε, κάναμε μία ευρωπαϊκή εκστρατεία κατά της ε, βίας ε, με βάση τη φιλοτική διάσταση. Κάναμε πολλές συζητήσεις σε επίπεδο επιτρόπων, χρηματοδοτήσαμε πάνω από 30 προγράμματα και έργα και διασφαλίσαμε την προσχώρηση στην ε, σύμβαση διασφαλίσαμε μάλλον την υπογραφή της ε, σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που είναι το πρώτο βήμα προς την ε, προσχώρηση. Είχαμε βέβαια και όλες αυτές τις αποκαλύψεις στο πλαίσιο του κινήματος MeToo που έδειξαν πόσο επίκαιρο είναι αυτό το ζήτημα και στην Ευρώπη. Κλείσαμε το έτος, τη χρονιά με, με μια εκδήλωση με ε, διεθνείς φορείς ε, που συμβάλλουν με μοναδικό τρόπο στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών ανά τον κόσμο. Επίσης, συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση ε, της διαδικασίας προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Παράλληλα, ασκούμε πιέσεις για την κύρωση της σύμβασης σε εθνικό επίπεδο. Σε ορισμένα κράτη-μέλη ε, έχει παρεμποδιστεί αυτή η διαδικασία για ιδεολογικούς και πολιτικούς λόγους που δεν συνδέονται με την ίδια τη σύμβαση. Συνεχίζουμε να προβάλλουμε ε, το μήνυμά μας και τη θέση μας και σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις για την κύρωση της ε, σύμβασης από πλευράς κρατών μελών και σας ευχαριστώ για την συνεχή σας στήριξη προς την Επιτροπή σε αυτό το σημαντικό φάκελο. Μπορώ να σας δώσω περισσότερες ε, λεπτομέρειες στη συνέχεια σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε με επιμέρους κράτη-μέλη και να, εδώ, να σας ζητήσω να μας βοηθήσετε γιατί πιστεύω ότι είναι ένας τρόπος να χειριστούμε καλύτερα ε, την κατάσταση αυτή αν και εσείς μας βοηθήσετε αν από κοινού προσπαθούσουμε να εξηγήσουμε στα κράτη-μέλη περί τίνος πρόκειται, γιατί κάποιες στιγμές ε, νομίζω ότι δαιμονοποιείται αυτή η σύμβαση, ενώ είναι μια πολύ χρήσιμη νομοθετική πράξη. Επίσης, ε, εκτιμώ ιδιαίτερα τη στήριξη της Επιτροπής ε, στην οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού βίου, ε, βασικό στόχο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, καθώς και βασική συνεισφορά στον εξυγχρονισμό της κοινωνίας μας. Το σχέδιο γνωμοδότηση που υποβάλλει σήμερα η κυρία Ράγεβιτς είναι μια εξαιρετική βάση ε, συζήτησης. Πρέπει να προχωρήσει αυτό ο φάκελο και να υιοθετηθεί εντός της κοινοβουλευτική αυτής Γιατί είναι κάτι απαραίτητο για τους πολίτες. Ε, να υπάρχει σημαντικό μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει βελτίωση τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό προσφέρουμε και στους άντρες και στις γυναίκες περισσότερες δυνατότητες να ε, συγκεράσουν ε, τις επαγγελματικέ και οικογενειακές τους υποχρεώσεις και ενθαρρύνουμε τον ε, ισομερή καταμερισμό των ευθυνών φροντίδας μεταξύ άντρων και γυναικών. Αυτή η ανάγκη αναγνωρίζεται όχι μόνο σε σχέση με τα παιδιά, αλλά και σε σχέση με άλλους συγγενείς που μπορεί να είναι εξαρτώμενα μέλη ή να είναι ασθενείς η καταβολή των επιμέρους ε, αδειών, ιδίως της βονικής άδειας, είναι από τις ε, πλέον καινοτόμε πτυχές της ε, οδηγίας. Είναι βασικό, βασικό στοιχείο για να υπάρχει σωμερής καταμερισμός στη φροντίδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αναμφίβολα, η νομοθετική μας πρόταση μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική σε συνδυασμό με αύξηση της διαθεσιμότητας προσιτή των εγκαταστάσεων ε, παιδικής μέρημνας. Η Επιτροπή ε, παροτρύνει τα κράτη-μέλη να αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους ε, προσφέρονται από τα διευθυντικά ταμεία για να επενδύσουν σε υποδομές φροντίδας. Και έχουμε, την, έχουμε σκοπό να δημοσιεύσουμε την επόμενη έκθεση αξιολόγηση για τους στόχους της Βαρκελόνης σε ό,τι αφορά την παιδική μέρημνα το Μάιο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ευρώπη κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι αρκετά γρήγορα. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος την κατάσταση των γεωνικών στην Ευρώπη με εσά, ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, ε, ηγετικέ φυσιογνωμίε από την κοινωνία των πολιτών, ακαδημαϊκού, νομικού, ακτιβιστέ, επιχειρηματίε και σωματεία, εκπροσώπους των μέσων ενημέρωση και δημοσιογράφου. στο ε, συνέδριο στο συμπόσιο του 2017 για τα θεμελιώδη δικαιώματα και διερευνήσαμε από κοινού τη σχέση μεταξύ τη ε, πλήρωση ε, και τη στήριξη του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων για τι γυναίκε και τον πλουραλισμό, την αλληλεγγύη, την ανοχή, ε, την ανεκτικότητα, δικαιοσύνη και την ισότητα. Και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να ενώσουμε τι δυνάμει μα και να αυξήσουμε τι προσπάθειε για να προαγάγουμε τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνήσαμε ότι αυτό πρέπει να γίνει και σε παγκόσμια κλίμακα με του ε, υπουργού ε, στο πλαίσιο του G7 το φθινόπωρο, όπου εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσίασα τι πολιτικέ μα. Μία από αυτές τις πολιτικές είναι η συμβολή μας για, την, ε, για τον περιορισμό του μισθολογικού χάσματος και ε, του συνταξιδοτικού χάσματος και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, επισημάνθηκε και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Πριν από αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος και θα υλοποιήσουμε τις 20 δράσεις στα επόμενα δύο χρόνια και επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή περαιτέρω συστάσεις στο πλαίσιο του Equality Bodies. Αυτή τη στιγμή ε, το Μάρτιο ε, έγινε ε, και το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ από την Βουλγαρική Προεδρία και πιο συγκεκριμένα μια συζήτηση για το κλείσιμο του μισθολογικού χάσματο μεταξύ των φίλων. Τα περισσότερα κράτη-μέλη τόνισαν την ανάγκη μια ολιστική προσέγγιση και συμφωνούμε, όμω ε, δεν πρέπει να μένουμε στα λόγια, χρειαζόμαστε πράξει. Γι' αυτό και έχουμε ε, την οδηγία ε, Women on Boards, αλλά και την οδηγία για τον για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού βίου και πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες δημοσιονομικές επιλογές. Όπως σημείωσα, Πρόσφατα τιμήσαμε την επέτειο της ε, παγκόσμια ημέρας της γυναίκας. Ε, επί, τη ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δημοσίευσε έκθεση για τις γυναίκες στον τομέα της πληροφορικής. Κάτι άλλο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε από συστημική άποψη και στηρίζω την ε, συνάδελφο Μαρία Γκάμπριελ ε, για να καταλήξει σε ένα ε, συνολικό σχέδιο για να διασφαλίσει την συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιοποίηση. Επίσης, συνεργάζομαι στενά με τη Σεσίλια Μάλστρομ σε ζητήματα που σχετίζονται με τις γυναίκες στο εμπόριο, αλλά και με την Βιολέτα Μπούλς για την ενσωμάτωση της φιλετικής διάστασης στις πολιτικές μεταφορών. Είδατε ότι στέκομαι ιδιαίτερα στη συνεργασία μου με τι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν όμω και άντρε. Ε, απλώς αυτά είναι τα τρία συγκεκριμένα παραδείγματα που ήθελα να σας αναφέρω. Από την έκθεση του 2018 για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία δημοσιεύσαμε την περασμένη εβδομάδα, είναι σαφέ ότι παρόλε τι ε, προσπάθειε και δεσμεύσει ε, να συνεχίσουμε σε αυτό το θεματολόγιο για την ισότητα των φύλων, είναι ε, πολύ μικρή η πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Και αυτό επιβεβαιώθηκε και από το Gender Equality Index που δημοσιεύσαμε το 2017 με το AGE και πραγματικά εκφράζω την απογοήτευσή μου, γιατί δεν βλέπουμε πρόοδο ή τέλο πάντων είναι πολύ μικρή η πρόοδο παρόλε τι ε, επενδύσει, δεσμεύσει και προσπάθειε που καταβάλουμε σε όλα τα δυνατά επίπεδα. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα ή κάτι δεν κάνουμε σωστά. Όμω πρέπει να το συζητήσουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν ε, συνεχή δέσμευση και προσήλωση από πλευρά μα. Σα ευχαριστώ όλους για την ε, στήριξή σας, ε, το έργο σας, την πολύ καλή συνεργασία και πάντα νιώθω ότι πραγματικά με στηρίζει αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στις εργασίες μας σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο, αλλά και στα επιμέρους κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την αγαστή συνεργασία και Είμαι πάντα στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επίτροπε για τα εισαγωγικά σας σχόλια και την ομιλία σας. Βεβαίως πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα εάν θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικά και θεαματικά αν θέλετε στην πράξη τα συμπεράσματα αυτών που θέλουμε να δούμε για την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε που ήρθατε εδώ ενώπιον αυτής της Επιτροπής. Είναι αλήθεια ότι εγώ συμφωνώ με την τελευταία σας σκέψη ότι έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε βέβαια και μου αρέσει να είμαι αισιόδοξη. Όμως ε, πρέπει να αναγνωρίσω ότι σε αυτή την ε, περίπτωση δεν ξέρω αν εξαρτάται από εμά ε, το αποτέλεσμα των όσων κάνουμε, γιατί κάναμε σχεδόν ολόκληρη τη θητεία μας με τσακωμούς, με προσπάθειες ευαισθητοποίησης για αυτό το θέμα και τα αποτελέσματα ήταν ισχνά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρώσουμε τα χέρια. Εγώ ως Ευρωπαίστρια και ως Φεμινίστρια ξέρω πάρα πολύ καλά πως πρόκειται για ένα διαρκή αγώνα, ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Και πρέπει βεβαίως ε, να συνεχίσουμε με κριτική ματιά για το τι γίνεται σε σχέση με την εργασία μας και τα αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να το κάνουμε με όλα αυτά τα θέματα που η δικιά μας Επίτροπος μας έχει βάλει επιτάπητος. Και ένας Ευρωπαίος πολίτης όταν τελειώσει αυτή η θητεία θα μας ρωτήσει ποια είναι τα επιτεύγματα που καταφέραμε ε, στο θέμα της ισότητας ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, εγώ θα δυσκολευτώ να απαντήσω. Θα μπορούσαμε να πούμε για τα όσα δουλέψαμε εδώ, για τα θέματα που μας απασχόλησαν, αλλά στην πραγματικότητα απλά, απτά αποτελέσματα τα οποία να μπορεί να τα αντιληφθεί ο Ευρωπαίος πολίτης ε, είναι περιορισμένα. Αρχίσαμε την θητεία διεκδικώντας την ανάγκη να αναθεωρηθεί η οδηγία για τις άδειες Μα Μας είπε η Κομισιόν ότι αξιολογούσε την νομοθετική δραστηριότητα και το καλύτερο να αποσύρουμε αυτή την πρόταση γιατί ήταν μπλοκαρισμένη στο Συμβούλιο και να υποβάλουμε νέα πρόταση. Κάναμε αυτή, έγινε αυτή τη δουλειά, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω, όμως ε, έχω σοβαρές αμφιβολίες, ε, δεν θα πρέπει, αν θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε πριν ολοκληρωθεί αυτή η θητεία, να προβούμε σε συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο, το, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για τις γονικές άδειες σε αυτή την οδηγία. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να σας ρωτήσω, εσείς τι αίσθηση έχετε από τις συνεδριάσεις που κάνατε με τους ηθήνοντες ε, ε, στο Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Θεωρείτε πως το Συμβούλιο θα, βρει, θα, θα, μας δώσει κάποια κοινή θέση που να διαπραγματευτούμε. Γιατί εμείς μπορεί να κάνουμε ό,τι θέλουμε στις συζητήσεις μας και στη δουλειά μας, αλλά ε, φοβούμε ότι μπορεί να συμβεί το ίδιο που συνέβη με την οδηγία για τις με, άδειες Δηλαδή το συζητήσαμε, εμείς καταλήξαμε σε κοινή θέση του Κοινοβουλίου και να μην χρησιμεύσει σε τίποτα γιατί δεν έχει βρεθεί κοινή θέση στο Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω αν υπάρχει, αν έχετε εσείς κάποιες περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτό το θέμα για το κατά πόσο θα ήταν βιώσιμο, τουλάχιστον να μπορούμε να ξεκινήσουμε του τριμερεί ε, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια θέση. Γιατί μπορεί να έχουμε διαφορές όσον αφορά το πώ πρέπει να είναι οι άδειε αυτές, ποιο θα τις πληρώνει, πόσο χρόνο θα είναι, αν θα μπορεί κανείς να τι μεταφέρει κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να βρούμε μια κοινή θέση που θα έχει την πλειοψηφία και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Τώρα, αν αυτή η θέση τελικά βρει μια μειοψηφία που θα την μπλοκάρει πάλι στο Συμβούλιο, θα είναι πάλι δύσκολο να το εξηγήσουμε στους πολίτες. Το ίδιο και με τη Σύμβαση της Ισταμπούλ, όπου γνωρίζετε, Επίτροπε, στην τελευταία ολομέλη έγινε συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα. Τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ, από αυτό το Κοινοβούλιο, που να μην το έχουμε κάνει ήδη. Θα μπορούσατε θα μπορούσαμε να, να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη επίμονα να την κυρώσουν. Το κάνουμε, αλλά φοβούμε ότι θα τελειώσει η θητεία και δεν θα έχει ολοκληρωθεί η από ευρωπαϊκής πλευράς η, η κύρωση αυτής της σύμβασης. Πώς θα εξηγήσουμε στους πολίτες τι έκανε αυτή η Κομισιόν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε θέματα ισότητας ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Ε, ε, δουλέψαμε. Ναι, εμείς εδώ στην Επιτροπή μας δουλέψαμε, επιμένω γι' αυτό. Και ε, θα πρέπει να σας αναγνωρίσουμε και τη δουλειά που κάνετε και εσείς ορισμένα από αυτά τα θέματα. Αλλά αν έχουμε ενώπιον μας, μάλλον απέναντί μα, ένα συμβούλιο το οποίο δεν είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις και δεν είναι σε θέση να μας καταλάβει για όλα αυτά τα σημαντικά θέματα, δυστυχώς θα πρέπει να είμαι εδώ απεσιόδοξη γιατί δεν βλέπω πολύ ρόδινο ε, το, το, τον ορίζοντα και το, την εικόνα μάλλον που, έχω, που δίνουμε. Εφόσον πρέπει να επικρίνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, αυτή είναι η δουλειά μας, ε, αυτή είναι το καθήκον μας ως βουλευτές και θα το κάνουμε, Επίτροπε, και σας ευχαριστώ. Και εγώ. Ευχαριστώ. Η Ντανιέλα Αγιούτα. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την Επίτροπο που είναι σήμερα παρούσα. Ήθελα εγώ να αναφέρω κάποια δύο θέματα διαφορετικά μεταξύ τους. Από τη μια πλευρά θέλω να σας μιλήσω για κάποια τελευταία γεγονότα περιστατικά. Το ένα μάλιστα συνέβη πριν από τέσσερις μέρες με διαφορετικό τέλος. Στα σύνορα της Γαλλίας με την Ιταλία αποθήθηκε μία γυναίκα που ήταν έγκυος και μετά από ε, λίγες ώρες πέθανε αφού ε, υπέστη κεσαρική τομή κατεπηγόντως. Απ' την άλλη είχαμε έναν οδηγό ε, της, ε, στα, ε, Γάλλο οδηγό στα βουνά ανάμεσα στην ε, Γαλλία και Ιταλία που έφερε τη γυναίκα, μια γυναίκα έγκυο που συνάντησε στο νοσοκομείο η οποία επέζησε και αυτός κατηγορείται τώρα ότι παράνομα έφερε μια πρόσφυγα μετανάστρια και κινδυνεύει να φυλακιστεί για πέντε χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε τελείως διαφορετικές περιστάσεις, όμως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η έλλειψη υποδοχής και πολιτικής υποδοχής κοινή ε, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα δεν ξέρω ξεκινήσουμε, δεν θέλω να ξεκινήσουμε με όλη συζήτηση που, για τα αίτια όλων αυτών. Πάντως τελικά αυτό που το πληρώνουν οι πιο αδύναμοι, όπως ε, οι γυναίκες δηλαδή, οι ε, μετανάστριες. Ρωτώ λοιπόν, ποια είναι η δική σας θέση για αυτά τα πολύ ε, διαφορετικά περιστατικά, αλλά και τι μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν για να μην ε, υπάρχουν τέτοια περιστατικά και έτσι ώστε οι γυναίκες να προστατεύονται καλύτερα και πιο συγκεκριμένα και να μην υπόκειται τις συνέπειες των πολιτικών και στρατηγικών σφαλμάτων που είναι τελείως διαφορετικής φύσης. Και το άλλο θέμα που θέλω να αναφέρω συνδέεται με την καταπολέμηση της βίας εναντίον στις γυναίκες και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι από το 1999 που δεν έχει γίνει ένα ευρωπαϊκό έτος ε, καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Τα τελευταία δύο χρόνια μάλιστα δεν υπήρξε καν ε, καμία πρωτοβουλία για αυτό το θέμα όπως έγινε για διάφορους άλλους ε, αγώνες και μάχες. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και πόσο η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού έτους για αυτό το θέμα μπορεί να συμβάλλει στο να συζητηθεί περισσότερο και στο να εφαρμοστούν διάφορες δράσεις στα διάφορα κρατή-μέλη που μπορεί να ευαισθητοποιήσουν, ας πούμε, για αυτό το θέμα δυστυχώς καθημερινά. Ε, βλέπουμε περιστατικά που, που, που μας θυμίζουν διαρκώς αυτό το θέμα και πραγματικά έχουμε κουραστεί να πρέπει να απαντάμε στους πολίτες και κυρίως στις γυναίκες πολίτες ότι ναι, ναι, υπάρχει νομοθεσία, κυρίως σε κάποια κράτη, ας πούμε στην Ιταλία, όπου υπάρχει νομοθεσία σχετική και καλή. Ωστόσο, δεν είμαστε ακόμα σε, θέμα, σε θέση να αποφύγουμε συγκεκριμένα περιστατικά. Άρα λοιπόν κάτι λείπει. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία λοιπόν που, μπορεί να αναλυφθεί, να αναλυφθεί. Δεν ξέρω αν έχετε προβλέψει κάτι και τι εμποδίζει τους θεσμούς ε, να θεσπίσουν ένα ευρωπαϊκό έτος ε, αφιερωμένο στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ευχαριστώ. Κυρία Σουντρόβα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. <coughs> Γιατί λόγια που μας είπατε. Θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά την κατάσταση στην Τσεχία, περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κάποια μέτρα δεσμευτικό χαρακτήρα όσον αφορά την ε, ισότητα των ε, ανδρών και γυναικών. Βεβαίως, πρόκειται για αρμοδιότητα εθνική είναι κάτι που θα πρέπει να το αναλάβουν τα κράτη-μέλη. Οι εθνικές αρχές είναι αυτές που είναι αρμόδιες. Όμως, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει ακριβώς ε, κάποια προετοιμασία με τις οδηγίες, με την απαγόρευση της νομοθεσίας αυτής που ε, ουσιαστικά οδηγεί σε διακριτική μεταχείριση και βλέπουμε ότι το να προσχωρήσουν στην ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι αποκλειστικά και μόνο αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η ίση μεταχείριση των γυναικών, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών επαναλαμβάνω, είναι κάτι που θα πρέπει βεβαίως να το αποφασίσουν και να το ελοπίσουν τα κράτη-μέλη. Αλλά μπορεί ένα είδος παρακολούθησης, monitoring να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν θέλουμε να συγκρίνουμε την κατάσταση από τη μία χώρα στην άλλη, για όλους αυτούς τους ομίλους μπορεί οποίους προαναφέρετε, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει κάτι. Να δείξει στα κράτη-μέλη πώς μπορούν να στηρίξουν και να συνοδεύσουν ε, τις γυναίκες σε αυτή την προσπάθειά τους για ίση μεταχείριση. Παραδείγματος χάρη, το θέμα της ε, επαγγελματικής ζωής και της ιδιωτικής ζωής, το θέμα της φροντίδας των παιδιών. Γνωρίζουμε τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι όσον αφορά όλον αυτό το τομέα τα πράγματα πάνε καλύτερα αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται μια έκκληση προς τα κράτη-μέλη για να υιοθετήσουν μέτρα στήριξης αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για τους άνδρες και τους γυναίκες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να γίνει παράδειγμα. Θα πρέπει να δράσει παραδειγματικά και να θέσει τον πύχη ψηλά θα πρέπει να βοηθήσει όλα τα κράτη-μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει μέχρι τώρα φιλόδοξα μέτρα για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και για τις ίσες ευκαιρίες που πρέπει να δίνονται στις γυναίκες να το κάνουν. Νομίζω ότι πραγματικά η παραδειγματική συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να εμπνεύσει και άλλα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εγώ θα ήθελα να σχολιάσετε, <clears throat> Επίτροπε, τι μέτρα θα προωθήσετε για αυτό το πακέτο ε, συνδιαλλαγής. Γιατί, ας πούμε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία έχουν ε, μπλοκάρει το θέμα. Και εγώ ρωτώ από αυτή την Επιτροπή, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, μπορούμε να επηρεάσουμε κάπου για να προχωρήσει αυτό το, αυτή η νομοθετική δέσμη για να μην μπλοκαριστεί πάλι από το Συμβούλιο αυτό το θέμα. Και δεύτερη ερώτηση, όσον αφορά τη Σύμβαση της Ισταμπούλ, τι να κάνουμε για να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να κυρώσουν και μάλιστα και να πείσουμε και αυτό το κράτος που έχει τώρα την Προεδρία. Και να σας θυμίσω γιατί ε, η Ισπανία ήταν μια από τις χώρες όπου υπήρξε τεράστια ε, κινητοποίηση γιατί ε, υπάρχει πρόβλημα με την βία κατά των γυναικών, πότε θα προωθηθεί αυτή η οδηγία για την καταπολέμηση της βίας ε, κατά των γυναικών, το φεμινιστικό κίνημα και όλες οι γυναίκες ε, στην Ευρώπη το ζητάμε και το είδατε και στις 8 Μαρτίου πως όντως το ζητάμε και μάλιστα πολύ έντονα. Ε, τίποτα άλλο, ευχαριστώ. Θα, θα είχα ακόμα ένα αίτημα. Το έχουμε ρωτήσει στην ήδη από την υπηρεσία της Ολομέλειας. Να ζητήσουμε δηλαδή ότι τα θέματα των δικαιωμάτων των γυναικών να μην μένουν τελευταίο στιγμή στην ημερήσια διάταξη, παρακαλώ. Ε, thank you very much. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε σήμερα εδώ, κύριε Επίτροπε, για άλλη μια φορά. Χαίρομαι που έχουμε αυτόν τον ε, συνεχή διάλογο μαζί σας. Και βεβαίως ε, από το 2014 έχουν προσυπογράψει όλα τα κράτη-μέλη για την πολιτική της ισότητας των φύλων. Όταν έχουμε όμως τεράστιες, αν θέλετε, διαδηλώσεις, όπως αυτό που έγινε στην Πολωνία, τη μαύρη διαδήλωση για την ε, αντίσταση κατά αυτής της ε, νομοθεσίας βλέπουμε ότι το θέμα των γυναικών πάντα βρίσκεται σε αυτές τις διαμαρτυρίες. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι το πιο αποτελεσματικό δεσμευτικά νομικό εργαλείο. Δεν καταλαβαίνω, είμαστε στο 1500, στο 1800, Είμαστε στο 1950 πριν γεννηθώ και αναρωτιόμαστε αυτό που αναρωτιόμαστε. Μα σήμερα όμως αυτό δεν είναι δυνατό τον 21ο αιώνα. Οι νέοι το έχουν καταλάβει. Έχουν καταλάβει τη σημασία του να υπάρχει πραγματική ισότητα των φίλων. Θα σας κάνω και μια άλλη ερώτηση διαφορετική. Το θέμα της ενσωμάτωσης καθώς και αυτά τα τρομακτικά πράγματα που συμβαίνουν κατά των ε, γυναικών. Ήμουν στη Βαρκελόνη την Παρασκευή και όλοι ξέρουν τι συμβαίνει με τις γυναίκες Ρωμά. Από τη στιγμή που ξεκίνησαν πάλι στην Ευρώπη εξτρεμιστικά, ρατσιστικά, νασιοναλιστικά κινήματα, βλέπουμε ότι το θέμα των μειονοτήτων, των γυναικών, στις μειονότητες επανήλθε στην καρδιά της ανησυχίας μας. Οι γυναίκες βεβαίως έχουν μία πάρα πολύ ισχυρή, αν θέλετε, αντιμετώπιση και αντίδραση. Όμως το θέμα της συμμετοχής στη δημόσια ζωή είναι κάτι που λείπει ακόμα. Θα ήθελα λοιπόν πάρα πολύ να σας μεταφέρω ένα μήνυμα από την ε, συνεδρία που ήμουνα. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε οι γυναίκες ε, που ανήκουν σε αυτές τις μειονότητες, οι γυναίκες μετανάστριες, ε, να βρεθούν πραγματικά σε μια κατάσταση με ίσες ευκαιρίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που για άλλη μια φορά ήρθατε στην ε, Επιτροπή μας. Πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση είμαστε ευγνώμονες γιατί μπορούμε για άλλη μια φορά να επανέλθουμε σε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μας, ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αλλά πριν από τρεις, τρία χρόνια, ήμουν εισηγήτρια για μια, μια έκθεση με ακριβώς αυτό το θέμα. Ποια ήταν τα συμπεράσματα της εργασίας μου τότε. Η Επιτροπή υιοθέτησε κάποια μέτρα, βεβαίως, που ήταν συνέπεια αυτής της προσπάθειας και μάλιστα Μιλήσαμε για κάποιους νέους ορισμούς, για μια περιγραφή πιο ουδέτερη κάποιων θέσεων. Μιλήσαμε για διαφάνεια, μιλήσαμε για αποδοχές, για κυρώσεις που ενδεχομένως θα έπρεπε να επιβάλλονται. Χωρίς κυρώσεις νομίζω δεν θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Μάλιστα είχαμε προτείνει στα πλαίσια της έκθεσής μου μία αν θέλετε απαγόρευση κάποιων διαγωνισμών, κάποιων ειτήσεων για υποβολή προσφορών, εάν δεν υπήρχε ίση δυνατότητα συμμετοχής άντρες και γυναίκες. Ερωτώ λοιπόν, έχουμε πλησιάσει σήμερα μετά από τρία χρόνια πιο πολύ προς μια πραγματική ισότητα ευκαιριών. Γιατί δεν έχει νόημα να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Εγώ από τότε που ανήκω σε αυτή την Επιτροπή, από το 2014, έχουμε υιοθετήσει ψηφίσματα, μιλάμε για ίσες αποδοχές, για τους άνδρες και τις γυναίκες. Δυστυχώς όμως δεν νομίζω ότι έχουμε πραγματική πρόεδρο. Η κυρία Ζωάννα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση για μας. Είναι καλό να τα συζητούμε όλα αυτά ευθέως. Έχετε δίκιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειωθεί νομοθετική πρόοδος και μάλιστα σημαντική. Δυστυχώς όμως στην πράξη δεν βλέπουμε ε, σημαντικά αποτελέσματα. Είναι οριακή μόνο πρόοδος. Ίσως κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά. Ίσως πρέπει να βγούμε έξω και να μιλήσουμε με γυναίκες έξω στον κόσμο, να δούμε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και από κοινού προσπαθήσουμε να βρούμε επικοδομητικές λύσεις που να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Και αυτό θα σημαίνει ότι οι προσπάθειές μας στο μέλλον θα μεταφραστούν σε πραγματική πρόοδο. Να επιστήσετε την προσοχή σας στις διαφορετικές νοοτροπίες και τρόπους σκέψης και να προτείνω δημόσιες εκστρατείες. Πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην αλλαγή της νοοτροπίας στο μέλλον, γιατί προς το παρόν περισσότερο το θέμα είναι οι επιλογές που έχουν οι γυναίκες. Όμως εγώ το έχω εξετάσει αυτό στη Ρουμανία. Έχω πάει και σε διασκέψεις για τι ε, ίσες ευκαιρίε, ε, για γυναίκε που εργάζονται σε συγκεκριμένου κλάδου, Έχω έρθει σε επαφή με πανεπιστήμια και στατιστικέ υπηρεσίε και είδα πόσε γυναίκε ουσιαστικά ε, ζητούν τεχνικές, ε, την αναγνώριση των τεχνικών τους προσόντων και δεν είναι πολλές. Και άλλα προβλήματα, μονογονικές οικογένειες. Εκεί πολύ συχνά οι γυναίκες μόνες τους φροντίζουν ένα, δύο, τρία παιδιά πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να στηρίξουμε αυτές τις γυναίκες, γιατί μιλούμε εδώ και για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού βίου, έτσι. Σας ρωτώ λοιπόν, πόση προσπάθεια θα πρέπει να περιμένουμε να καταβάλει μια γυναίκα στην καθημερινότητά της. Κάποιες φορές αυτές οι γυναίκες καταβάλουν τη διπλή και τριπλή προσπάθεια σχέση με άλλους, γιατί και δουλεύουν για δουλειές και έχουν και δύο-τρία παιδιά και πρέπει να τα φροντίσουν στις μονογονικές οικογένειες αναφέρομαι. Η γυναίκα λοιπόν δεν έχει κάποιον να φροντίσει ε, τα παιδιά της όταν εκείνη εργάζεται. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερα ε, για να τις βοηθήσουμε στην πράξη με πρακτικές λύσεις λοιπόν. Μίλησα πριν και για τις ε, δημόσιες εκστρατείε, Πρέπει να έχουμε τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης για να υπάρχει πραγματική ισορροπία μεταξύ προσωπικού και, και προσωπικού χρόνου. Πρέπει να αλλάξουν η νοοτροπία μας λοιπόν. Σημαντικό εδώ είναι και η κατάσταση των γυναικών στην Ήπεθρο. Μιλούμε για ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα, αλλά τι γίνεται με τις γυναίκες που ζουν στην Ήπεθρο, ε, μακριά τα αστικά κέντρα, δεν έχουν ε, ε, πώς, τρεχούμενο νερό, δεν έχουν άλλες υποδομές δεν υπάρχουν δημόσιες συγκοινωνίες για να πάνε εκείνοι στα παιδιά τους, στην πόλη, να πάνε στη δουλειά, στο σχολείο. Ε, καλή λοιπόν η συζήτηση για τις ίσες ευκαιρίε, αλλά δεν πρέπει να μιλούμε μόνο για τα αστικά κέντρα, πρέπει να μιλήσουμε και για την Ήπεθρο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι δεν γίνεται να το συζητούμε μόνο στην Επιτροπή ΦΕΜ πρέπει να ασχοληθούν με αυτά τα ζητήματα όλε οι αρμόδιες επιτροπέ, περιφερειακή ανάπτυξης, γεωργίας, ίσως και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Όλοι από κοινού λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις για αυτά τα κοινά προβλήματα. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που υπάγονται στις δικέ μας αρμοδιότητες. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα ε, επιδόματα για όσου έχουν παιδιά αλλάζουν αυτά από χώρα σε χώρα, αλλά έχουμε να κάνουμε εδώ με τα δικαιώματα των γυναικών και πρέπει να, να εξετάζουμε και τα δικαιώματα των παιδιών τους. Προτείνω λοιπόν το εξή. Να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εξίσωσης ε, των ε, επιδομάτων, ίσως ένα καταποκοπήν επίδομα να υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη, ε, το ίδιο δηλαδή, για να στηρίξουμε και τις αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν δώσουμε ίση ε, στήριξη και ίσα επιδόματα σε όλα τα κρατημέλα, εξάρτητα το που μένει κανεί. Η κυρία Κοσλόσκα τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα. Δυστυχώ δεν ήμουν εδώ το πρωί, ε, συγγνώμη, στην αρχή τη συνεδρία, γιατί έπρεπε να ψηφίσω αλλού. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τις ε, προλαλήσασες ότι ο κατάλογος των αρμοδιοτήτων είναι ιδιαίτερα μακροσκελής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι είναι ε, ε, το φόρουμ που προβάλλει περισσότερο αυτήν, αυτόν τον τομέα πολιτικής και όπως συχνά έχουμε νέες νομοθετικές προτάσεις, όμως παραμένουν ορισμένες αφιβολίες. Η αδυναμία είναι κατά πόσο όλα αυτά που συζητούμε και αποφασίζουμε εδώ εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ για την δέσμη μέτρων ε, εξισορρόπησης επαγγελματικού και προσωπικού βίου. Περιέχει καλές προτάσεις, όμως κυρίως πρέπει να μεριμνήσετε για την ε, ε, προώθηση αυτής της ε, πρότασης στην πράξη και την ολοποίηση της στην πράξη. Νομίζω ότι για πρώτη φορά ε, υιοθετείται νομοθεσία για τις γυναίκες στον επαγγελματικό χώρο και δεν κάνει λόγο, δεν επικαλείται μόνο τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και την ισότητα μεταξύ άνδρων και γυναικών. Αυτή είναι η βασική μας ε, αρχή λοιπόν. Δεύτερον, αυτή η νομοθεσία είναι σημαντική γιατί δίνει τη δυνατότητα πραγματικής σύνδεσης μεταξύ ε, του επαγγελματικού και προσωπικού βίου. Γιατί και, τα δύο, ε, και στα δύο μέρη εργάζεται κανείς, και στη δουλειά του και στο σπίτι. είναι διαφορετικές μορφές εργασίας. Υπάρχουν και πολλές γυναίκες ε, που δουλεύουν από το σπίτι, αλλά για παράδειγμα όταν αρρωστήσει το παιδί τους, τι να κάνει μια τέτοια γυναίκα. Πρέπει λοιπόν σε μια τέτοια πρόταση να, διασφαλίσουμε μια πραγματική ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού βίου και εργασίας στο σπίτι. Και χαίρομαι που κάνετε αυτή την ε, πρόταση και η πρόταση ε, για την ε, φροντίδα γιατί μεγάλο τμήμα της φροντίδας για ένα παιδί λαμβάνει χώρα στο σπίτι. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν ε, υποδομές μέρημνας για τα παιδιά, παιδική σταθμή και το καθεξής, όμως μεγάλο τμήμα της φροντίδας παιδιών γίνεται στο σπίτι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση. Και ελπίζω και αυτοί και άλλες προτάσεις που θα εξετάσουμε στο μέλλον θα εστιάζουν την προσοχή πραγματικά στην εφαρμογή, στην υλοποίηση αυτής της νομοθεσίας. Γιατί τι να την κάνουμε την καλύτερη νομοθεσία αν δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε το λόγο στην Επίτροπο για να απαντήσει. Ακούσατε πολλά ερωτήματα. Έχουμε 15 λεπτά. είναι όχι τόσο ερωτήσεις, είναι και πολύ σημαντικές ε, ε, και επικοδομητικές οι προτάσεις και οι ιδέες σας, γιατί πραγματικά εμπλουτίζουν αυτό το διάλογο. Πρώτα απ' όλα, για αυτά που είπε η κυρία Γαρθία Πέρεθ. Νομίζω ότι ε, και εγώ προβληματίζομαι και εκνευρίζομαι γιατί δεν βλέπω τις ίδιες, την πρόοδο που θέλαμε και αυτό είναι απογοητευτικό. Πρέπει όμως να εκτιμήσουμε και τη διαδικασία, όχι μόνο την επίτευξη στόχων. Δείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Βέβαια, σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχει πισωγύρισμα, σίγουρα. Οπότε εκεί ε, εξυμνούνται τα παραδοσιακά οικογενειακά πρότυπα. Άκουσα πρόσφατα ότι πρέπει να καταλάβει η γυναίκα ότι ε, ανήκει στην κουζίνα. Πραγματικά δεν περίμενα να το ακούσω αυτό από κάποιον που έχει εκλεγεί. Και δεν τα έλεγε βέβαια τόσο ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά δεν έκρυψε την οτροπία του αυτή μετά. Ε, προάγει αυτές τις ε, ιδέες και εξελέγει αυτό που είπε η κυρία Σόιντροβα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι η πιο ισχυρή φωνή που θα προάγει αυτές τις αξίες. Και θα εξακολουθήσει να προάγει αυτή την πολιτική, γιατί στα κράτη-μέλη μπορεί να υπάρχουν εξελίξει που θα μα εκπλήξουν, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σταθερή. Αναφέρατε την ε, μαύρη διαδήλωση στην ε, Πολωνία. Ε, Ήρθα στο Κοινοβούλιο φορώντα μαύρα, ντυμένη στα μαύρα και με κατηγόρησαν ότι δεν είμαι ουδέτερη, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Μα πώ γίνεται ω γυναίκα να μείνω ουδέτερη σαφώς και παίρνω θέση και ως γυναίκα και ως επίτροπος. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει θέση και να επιμείνει σε αυτή τη θέση. Πρέπει λοιπόν να το εκτιμήσουμε αυτό σαν διαδικασία. Κάποιες φορές με απογοητεύει το γεγονός ότι λέμε πολλά, αλλά τελικά κάνουμε λίγα. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα συνομίλησα και συζήτησα με του υπουργού το μισθολογικό χάσμα και είπαν ότι ε, έχουμε πρόβλημα, αλλά δεν ακούμε κάποια λύση. Δεν έχουν γίνει ορατές ε, οι λύσεις. Τα απτά αποτελέσματα είναι τα νομοθετήματα και συμφωνώ με την τελευταία ομιλήτρια ότι η εφαρμογή είναι ζωτική σημασίας. γιατί επενδύουμε πόρους στις εκστρατείες, στηρίζουμε ε, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, εργαζόμαστε σε πολλά μέτωπα και μπορεί να μην είναι τόσο ορατά αυτά τα αποτελέσματα, αλλά είναι υπαρκτά. Θα ήθελα να τονίσω ε, θα πρέπει να είναι αμφίδρομη αυτή η διαδικασία και εμεί ω πολιτικοί θα πρέπει να λειτουργήσουμε και να δράσουμε από τα πάνω, αλλά πρέπει να υπάρχει και απαραίτητη βούληση σε κοινωνικό επίπεδο. Οι γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες, για παράδειγμα, πρέπει και αυτές ε, να ε, αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, γιατί πολλές γυναίκες ε, διαμαρτύρονται ότι είναι δύσκολη ζωή τους, πρέπει να έχουν πολλές ε, ε, ευθύνες, πολλές δουλειές να κάνουν σε πολλά μέτωπα, αλλά παράλληλα λένε ότι πρέπει, θέλουν να διατηρήσουν τη ζωή όπως, όπως την έχουν μάθει. Γιατί στατιστικά βλέπουμε ότι αυτές οι γυναίκες δυσκολεύονται, αλλά λένε ότι δεν θέλουν τις αλλαγές. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου και αυτό, ότι σε ορισμένες κοινωνικές κατηγορίες οι γυναίκες δεν επιθυμούν αυτές τις αλλαγές. Οπότε θα είναι πιο δύσκολο να αλλάξουμε τα πράγματα εκεί και θα μας πάρει περισσότερο καιρό. Τώρα πιο συγκεκριμένα. Ναι, αποσύραμε την οδηγία για την ε, άδεια μητρότητα και υποσχεθήκαμε να το αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο. Είναι λοιπόν η δέσμη για την ισορροπία προσωπικού και επαγγελματικού βίου στα μη νομοθετικά. Η κυρία Γκαρσία Πέρες ρώτησε τι συμβαίνει στο Συμβούλιο. Να σας πω θέλουμε να πετύχουμε γενική προσέγγιση την 21η Ιουνίου. Χλώμιασε η συνάδελφος, γιατί είναι υπέρ, αρμοδια αυτά τα ζητήματα. Όμως ε, νομίζω ότι μπορούμε να τα, καταφέρουμε εάν υπάρξει πνεύμα συμβιβασμού και από ε, το Συμβούλιο εγώ θα πω σίγουρο ότι είμαστε ανοιχτοί στο συμβιβασμό, αρκεί να μην ε, ακυρώνουμε τον σκοπό των οδηγιών, έτσι. Ορισμένα κράτη-μέλη ε, διαφωνούν με τους τέσσερις μήνες, θέλουν να πάμε στους δύο μήνες. Δεν είναι βέβαια το ιδανικό αυτό, για να πω και εγώ την γνώμη της Επιτροπής. Κάποιοι δεν ε, θέλουν αυτόν τον ορισμό της άδειας ασθένειας, sick pay, γιατί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δεν ασχολείται με αυτή την, δεν λειτουργεί με αυτή την κατηγορία ε, πληρωμών. Έχει διαφορετικό σύστημα λοιπόν. Μπαίνουμε δηλαδή στο, ε, στο επιμέρους ε, σύστημα τη κάθε χώρα όπου υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα και δυσκολίε. Πρέπει λοιπόν και εδώ να καταλήξουμε σε μια σημαντική πρόταση, να βρούμε τη διατύπωση που ε, θα εξυπηρετεί το σκοπό που θέλουμε, δηλαδή να υπάρχει οικονομική στήριξη προς ε, του εργαζόμενου γονεί, αλλά να είναι και κάτι εφαρμόσιμο από τα κράτη-μέλη. Για τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το πιο δύσκολο μάλλον προ το παρόν. Κάποια κράτη-μέλη διαφωνούν με τα 12 έτη ηλικίας ε, του παιδιού. Υπάρχουν πολλές πιέσεις από τις ενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί λένε ότι αν ε, αναλάβουμε εμεί όλο το βάρος, ε, τότε αυτό θα μας καταστρέψει. Και θα έχει πολύ σημαντικές επιπλοκές για εμάς. Για πολλούς λόγους, δεν έχω αρκετό χρόνο να τα αναλύσω. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει έδαφος λογικών συμβιβασμών και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για να πετύχουμε γενική προσέγγιση μέχρι τις 21 Ιουνίου. Θα ήθελα να ολοκληρωθεί και να ε, υιοθετηθεί μέχρι το τέλος της θητείας μας, γιατί πιστεύω ότι αυτό το ένα σύνολο νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων μπορεί να οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα. Και βέβαια έχουμε να κάνουμε και με το μεγάλο ε, ζήτημα που αντικατοπτρίζεται στη δέσμη για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού βίου και νομίζω ότι η Επιτροπή έκανε πλήρη μεταβολή. Ε, εγώ έστειλα επιστολή σε όλες τις ε, σχετικές υπηρεσίες για ανακατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ανάπτυξη των υπηρεσιών που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και προσιτές ε, στους εργαζόμενους γονείς και στις ε, γυναίκες, ε, στις μονογονεϊκές οικογένειες. Γιατί εδώ αυτό άπτεται άμεσα της φτώχειας. Είναι λοιπόν πραγματικά απαραίτητο να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτές τις γυναίκες που μεγαλώνουν μόνο τα παιδιά τους για να καταφέρουν να επιβιώσουν. για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Αυτό με φέρνει σε αμηχανία, γιατί ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να έχουμε ώστε να το περισσότερες αρμοδιότητες αλλά η διαδικασία οδηγεί τελικά στον περιορισμό των αρμοδιοτήτων μόνο στις αποκλειστικές αρμοδιότητες που μας ε, εκχωρεί η συνθήκη. Έχουμε σοβαρά προβλήματα σε μια σειρά κρατών μελών, Ακόμα 11 κράτη-μέλη δεν έχουν ε, κυρώσει τη σύμβαση και σε ορισμένα κράτη-μέλη από ό,τι φαίνεται υπάρχει ιδεολογικό ζήτημα και εγώ δεν το κατανοώ γιατί αυτό έχει να κάνει με την υγεία και τη ζωή γυναικών και παιδιών. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω ότι στο καλό είναι ιδεολογικό σε αυτή τη συζήτηση, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τα επιχειρήματα που ακούω κάποιες φορές. Η μεθοδολογία που βάζουν από το παράθυρο για το τρίτο φύλλο λένε ότι εμείς επιβάλλουμε με το ζόρι την σεξουαλική αγωγή στα σχολεία και το καθεξής. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τρία είναι λοιπόν τα προβλήματα. Γλωσσικό ζήτημα, σε κάποιες γλώσσες δεν υπάρχει διαφορετική, διαφορετικός όρος για το sex and gender. Αυτό είναι μια πραγματική δυσκολία γιατί έχουν διαφορετικό νόημα αυτές οι δύο λέξεις. Μετά και σε κάποιες μεταφράσεις αν δεν μεταφραστεί σωστά η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ε, παρερμηνίες και έχουμε κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για να το διορθώσουμε. Και τέλος ε, υπάρχει και σκόπιμη παρερμηνία της σύμβασης για ιδεολογικούς λόγους. Και σε μια παραδοσιακή οικογένεια. Εγώ πάντα υπερασπίζομαι την οικογένεια, αλλά τώρα για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο παραδοσιακή οικογένεια, Εμεί δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Η παραδοσιακή οικογένεια μπορεί να είναι και αυτή στην οποία υφίστανται κακοποίηση η γυναίκα και τα παιδιά δεν πρόκειται να το αφήσω έτσι. Θα πάω σε αυτά τα κράτη-μέλη ε, με βάση και τι δεσμεύσει δεσμεύσεις μου μέχρι τα τέλη Μαΐου. Λοιπόν, θα μεταβώ σε αυτά τα κράτη-μέλη και θα συμμετάσχω προσωπικά στην εκστρατεία για τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολης. Αν μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε στα κράτη-μέλη, ε, παρακαλώ να το κάνετε πραγματικά. Θα σας πω ποια είναι τα κράτη-μέλη στα οποία έχουμε δυσκολίες. Βουλγαρία, Σλοβακία, Λετωνία και Κροατία προς το παρόν. Νομίζω ότι και στη δική μου χώρα θα υπάρξει ζωηρή συζήτηση. Η συνάδελφος λοιπόν ε, και ε, συμπατριώτησά μου μπορεί να με βοηθήσει. Πραγματικά δεν περίμενα να πάρουν τέτοια τροπή συζητήσει. Ήλπιζα ότι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα γίνει κατανοητή ως αυτό που είναι, ένα πολύ χρήσιμο νομοθέτημα που δίνει αποτελεσματικές λύσεις για την κατηπολέμηση της βίας. Όμως δυστυχώς δεν ε, έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλουμε. Η κυρία Γιούτα. Θα εξετάσω αυτές τις ε, υποθέσεις φυσικά. Δεν μπορώ τώρα να υπησέλθω σε λεπτομέρειες, μπορώ όμως να ρωτήσω ποιες είναι οι ενέργειες των ε, αρμόδιων φορέων. Ξέρετε ότι προτεραιότητα ε, της Επιτροπής είναι η υιοθέτηση της νομοθεσίας. Οπότε σίγουρα υπάρχει ένομα ενδιαφέρον και ε, μπορώ να προσπαθήσω να ε, ρωτήσω πώς εφαρμόστηκε αυτή η οδηγία για την προστασία των γυναικών. Και μετά έχουμε και τους κανόνες για την ειδική μεταχείριση των ευάλωτων πολιτών. Για τις εγγύου, για παράδειγμα, σίγουρα υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία. Έχουμε ειδικού κανόνες για αυτές τις κοινωνικές ομάδες, ε, για πρόσφυγες και μετανάστες επίσης. Υπάρχει λοιπόν ένα σύνολο συγκεκριμένων ε, προϋποθέσεων που θα πρέπει να γίνεται σεβαστό. Θα το εξετάσω λοιπόν, δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι κάτι θα αλλάξει, αλλά θα του δώσω τη ιδέουσα σημασία. Μπορούν να αποτελέσουν βέβαια αυτές τις υποθέσεις προηγούμενο και να τα χρησιμοποιήσω στη συζήτησή μου με τα κράτη-μέλη που μας δημιουργούν δυσκολίες για να μην επαναληφθούν αυτά τα φαινόμενα. Για τη βία κατά των γυναικών, πέρσι είχαμε το ένα έτος που το αφιερώσαμε σε μία σειρά δράσεων. Είχαμε την εκστρατεία, είχαμε το συμπόσιο. Ακόμα χρηματοδοτούμε 30 προγράμματα στα κράτη-μέλη σε διάφορους τομείς που απευθύνονται κυρίως στους άνδρες και στα αγόρια. Ε, στην Ιταλία υπάρχει ένα πολύ καλό, ε, μια πολύ καλή καμπάνια ε, για τις ποδοσφαιρικές ομάδες. αλλά και στον κινηματογράφο έχουμε επενδύσει ένα ευρύ φάσμα λοιπόν ενεργειών που αναλάβαμε πέρσι. Πολλοί από σας θέλατε να αφιερωθεί αυτό το έτος στην καταπολέμηση της βίας και το πράξαμε. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά γιατί βέβαια το φαινόμενο δεν έχει εξαλειφθεί ακόμα. Πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν περισσότερα κονδύλια και προσπάθειες. Και ε, σε πρακτικό επίπεδο δεν υπάρχουν αρκετά καταφύγια για παράδειγμα κέντρα υποδοχή ε, αυτών των κακοποιημένων γυναικών. Υπάρχουν τέτοια κενά ε, και χρηματοδοτικά. Πρέπει να βρούμε τρόπο να στηρίξουμε ε, αυτές τις δραστηριότητε. Αυτό είναι καθήκον για μένα και στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, γιατί τώρα εξετάζουμε την περίοδο μετά το 2021. Αν δεν καταφέρουμε λοιπόν να εντάξουμε αυτή την πολιτική στο ευρύτερο ΠΔΠ, θα αποτύχουμε για τα επόμενα 7 χρόνια. Και σε αυτό μπορείτε να βοηθήσετε. Περιμένω λοιπόν να ακούσω και τις δικές σας προτάσεις ε, εκεί που εντοπίζετε ότι πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση. Φυσικά γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ του soft financing ε, που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε απευθείας από, τα, το πρόγραμμα δικαιοσύνης μας, αλλά υπάρχουν πολλά τέτοια κονδύλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στα κράτη-μέλη, που και αυτά θα πρέπει να αξιοποιηθούν ήδη από τώρα αλλά και για τον ε, επόμενο προπολογισμό θα υπάρχουν σημαντικά κονδύλια για τους, πόρους, για τους στόχους μας. Ε, λόγος γίνεται και για τα επενδυτικά κονδύλια, για παράδειγμα για τα καταφύγια αυτά και για τις ε, εγκαταστάσεις παιδικής μέρημνας. Κυρία Ιούτα, Νταϊούτο μάλλον, πράγματι είναι ελλειπής η εφαρμογή του νόμου. Συμφωνώ, πρέπει να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση για την εφαρμογή. Κυρία Σόιντροβα, είπα και εγώ πριν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκπληρώσει αυτό το καθήκον, να σηκώσει ψηλά ε, τη σημαία και να μην κάνει βήμα πίσω στην πρόθεση αυτών των ε, αξιών. Είναι θέμα αυτό κατά τη γνώμη μου. Πρέπει λοιπόν ε, να είμαστε απολύτως αμετακίνητοι σε ό,τι αφορά την ισότητα των, και ανυποχώρηση σε ό,τι αφορά την ισότητα των ε, φίλων. Βέβαια, απαιτείται αυτή η αμφίδρομη διαδικασία. Υπάρχει και το πολιτικό καθήκον, αλλά και το κοινωνικό καθήκον. Από κάτω προς τα πάνω ε, πρέπει να λειτουργήσουν ε, αυτές οι διαδικασίες. Και μπορεί να υπάρχουν ορισμένες ευβολίες κατά πόσο, για παράδειγμα, όσοι κατηγορούνται για σεξουαλική παρανόχληση είχαν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον αυτόν του. Πρέπει να το δούμε και από αυτή την άποψη. Αλλά αυτή η εκστρατεία, οι γυναίκες ε, στους δρόμους των Βρυξελών, της ε, Μαδρίτης, ανοίγουν τα μάτια ε, του κόσμου. Βλέπει ο κόσμος ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή εδώ. Και εγώ δεν λέω ότι ο κόσμος πρέπει να βγει στους δρόμους, αλλά αυτή είναι και η ομορφιά της δημοκρατίας, της δημοκρατικής κοινωνίας. Και επί τη ευκαιρία, δημοκρατικές κοινωνίες και εκστρατείες. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά ασχολούμαι πολύ με το ε, σκάνδαλο του Facebook. Γιατί εδώ είναι σοβαρή υπόθεση. Μια εταιρεία συλλέγει τα δεδομένα σου, φτιάχνει ένα προφίλ για σένα και σε βάζει σε μια κατηγορία βάση του αλγόριθμου και σε χειραγωγεί πλήρως σε ό,τι αφορά <laughs> την εκλογική σου στάση και τις πολιτικές σου αποφάσεις. Μπορεί να μην φαίνεται τόσο συναφές με αυτό που εξετάζουμε σήμερα. Πιστέψτε με όμως, έχει πολύ μεγάλη σχέση. Γιατί αν στο μέλλον διατηρηθεί αυτή η πρακτική, μπορεί όσοι υπερασπίζονται αυτές τις ε, παλιές παραδόσεις να κερδίζουν όλα και περισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις και νομίζω ότι εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να προστατεύσουμε τις ε, θεμελιώδεις μας ε, αξίες, όχι μόνο την εκλογική ελευθερία και την ελευθερία του ατόμου να επιλέγει ελεύθερα, αλλά και για την ισότητα στην κοινωνία, την αποφυγή των διακρίσεων και μια σειρά άλλα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό λοιπόν αυτό, πρέπει να το διερευνήσουμε όχι μόνο από πλευράς προστασία δεδομένων, γιατί αυτό είναι πολύ απλό. Έχουμε κανόνες και κυρώσεις για όσους τους παραβιάζουν, αλλά αυτό είναι πολύ ε, σοβαρό. Θα αναλύσουμε τη σοβαρότητα του φαινομένου και σε ό,τι αφορά την ε, ε, επιρροή που ασκείται στις δημοκρατικές διαδικασίες και θα εξετάσω πιο συγκεκριμένα και το θέμα των διακρίσεων γιατί νομίζω ότι απαιτούνται ενέργειες. Αυτό αφορά και συνδέεται και με το θέμα των γυναικών στην ψηφιακή εποχή που κάποιοι αναφέρατε. Θα επανέλθω προς την κυρία Σόιντροβα. Ναι, πρέπει όντως να κάνουμε το benchmarking. Ε, πολύ σημαντικά όλα αυτά. Υπάρχει και το ευρωβαρόμετρο, έχουμε νέα δεδομένα για την αντίληψη σε ό,τι αφορά την βία κατά των γυναικών σε ορισμένα κρατημέλη και σε σχέση με το πόση ανοχή υπάρχει απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Είναι ε, ενδιαφέρον ο σχετισμός αυτός μεταξύ ανοχής στην κοινωνία και ε, βίας. Βεβαίως υπάρχουν ακόμα μισθολογικές διαφορές ε, και διαφορετική επαγγελματική μεταχείριση. Κυρία Ταλάνοβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε αυτή την ερώτηση. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Μιλήσατε και για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Πού είστε όμως. Ναι, σας είδα. Εγώ κάνω μια έκκληση προς όλους σας. Αν θέλετε αν θέλετε, περισσότερα στοιχεία για το πώς η κάθε χώρα, η συγκεκριμένη δική σας χώρα, τηρεί, σέβεται την ίση εκπροσώπηση και μεταχείριση των ανδρών και γυναικών, μπορούμε να σας δώσουμε αυτά τα στοιχεία. Συμφωνώ επίσης ότι οι γυναίκες πλήττονται διπλά. Προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε με κοινοτική χρηματοδότηση με το κοινό πρόγραμμα παραδείγματο χάρη της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις γυναίκες Ρωμά και την πρόσβασή τους στην ε, δικαιοσύνη. Η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ρουμανία ε, έχουν υποφεληθεί ε, από το πρόγραμμα αυτό μέχρι τώρα. Πολλά προγράμματα όμως ε, αφορούν τους Ρωμά και ειδικότερα τις ε, γυναίκες Ρωμά και χρειάζεται μεγάλη, αν θέλετε, δουλειά όχι μόνο για τις γυναίκες Ρωμά αλλά και για τα παιδιά, ο αναλφαβητισμός, τα προβλήματα στον τομέα της παιδείας, κάτι που έχει άμεση σχέση βέβαια και με τις γυναίκες, με τις μητέρες. Στην ε, Βουλγαρία είδα ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα για καλύτερη πρόσβαση των ε, γυναικών Ρωμά στις υπηρεσίες υγείας. Αλλά αν σας ενδιαφέρει έχω πολλές πληροφορίες και μπορώ να σας τις ε, δώσω. Κυρία Ζαμπόρσκα, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που αναφέρατε, για αυτήν την δράση στην οποία συμμετέχετε και βεβαίως ε, το θέμα των κυρώσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό. Χωρίς κυρώσεις δεν υπάρχει αποτελεσματική δράση. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πρέπει να υποβάλουμε τροπολογίες που θα προτείνουν από τη μία κυρώσεις και από την άλλη υποχρέωση διαφάνειας. Ζητάμε διαφάνεια από μέρους των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα δεν είναι μέχρι τώρα πολύ ικανοποιητικά. Χρειάζεται, αν θέλετε, συμπλήρωμα και ελπίζω όταν ολοκληρωθεί η δική μου θητεία ο διάδοχός μου θα μπορέσει να βασιστεί σε αυτά που κάναμε και να κάνει αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμα συμπληρωματικά. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη όπου αν είσαι γυναίκα και διαπιστώσεις ότι πληρώνεσαι λιγότερο από τον ε, συνάδελφό σου που είναι άντρας και δεν έχει τη δυνατότητα και τα οικονομικά μέσα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, εκεί η κατάσταση είναι απογοητευτική και οι γυναίκες δεν διαθέτουν δυνατότητες να αμυνθούν και να αντισταθούν σε αυτό. Γι' αυτό και μιλήσαμε και για την ε, αστυνομία για θέματα ισότητας. Θα πρέπει εκεί να μπορεί να προσφύγουν οι γυναίκες δωρεάν όταν υπάρχουν τέτοιου είδους ε, μισθολογικές διαφορές, παραδείγματο χάρη. Αστυνομία για θέματα ισότητας και δικαιοσύνης και δίκαιης εκπροσώπησης των φύλων. Είναι κάτι που σας ε, υπόσχομαι ότι θα περάσει από soft law σε hard law, θα γίνει δηλαδή νομοθεσία. Ακούσαμε και κάτι άλλο που αφορά την διαφορά αποδοχών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το πιο σημαντικό είναι ότι κάποιες κατηγορίες με επαγγελματικές, κάποιες θέσεις απασχόλησης ε, με υψηλές αποδοχές ουσιαστικά δεν αφορούν τις γυναίκες. Ελάχιστα κορίτσια βρίσκονται εκεί. Οι γυναίκες βρίσκονται μαζικά και κατά κύριο λόγο στα επαγγέλματα αυτά τα οποία δεν αμείβονται καλά. Και εδώ για να πετύχουμε δικαιοσύνη και ίση εκπροσώπηση πολλά πρέπει να γίνουν. Ο δρόμος είναι μακρύς. Κυρία Ζωάννα, μιλήσατε για τις δημόσιες εκστρατείες και μιλήσαμε και για τον ψηφιακό κόσμο. Εγώ σας είπα πόσο με απασχολεί αυτό τον καιρό το σκάνδαλο με το Facebook. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να έχουμε μια προληπτική δράση, να λάβουμε μέτρα πρόληψης. Δεν υπάρχει αρκετός ε, αριθμός γυναικών ούτε στα μέσα, ούτε στον ψηφιακό κόσμο, ούτε σε υψηλόβαθμες θέσεις που επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ψηφιακή οικονομία, η τεχνητή νοημοσύνη, δύο εξαιρετικά σημαντικοί τομείς στους οποίους θα πρέπει οι γυναίκες να δραστηριοποιηθούν είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. Αν οι γυναίκες δεν μπουν σε αυτούς τους τομείς, θα χάσουμε άλλη μια ευκαιρία και θα είναι τρομακτική η αποτυχία και για τις γυναίκες και για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ε, αναπηρίες. Πολύ φοβάμαι, και αυτό είναι πολύ δύσκολο για μένα να το εκφράσω έτσι, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τα άτομα με αναπηρίες και οι γυναίκες θα βρεθούν σε μια κοινή κατηγορία εάν χάσουν το τρένο της ψηφιακής επανάστασης. Οι γυναίκες ε, στην Ήπεθρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ εμπνευσμένη ιδέα σας. Πολύ σύντομα θα βρεθώ στην ε, Επιτροπή των Περιφερειών και θα μιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Όπως σας είπα πρέπει εδώ να στοχεύσουμε το νέο προϋπολογισμό και δεν πρέπει να χάσουμε και αυτή την ευκαιρία να κατευθύνουμε καλύτερα τα πράγματα με τα μέσα που μας προσφέρει ο νέος προϋπολογισμός. Κυρία Κοσλόφσκα, νομίζω ότι απάντησα σε αυτό που μου είπατε, αλλά σας ευχαριστώ γιατί μιλήσατε για την ε, μερική απασχόληση και τις παγίδες. Έχετε δίκιο. Από τη στιγμή που οι γυναίκες μπουν στην κατηγορία της μερικής λεγόμενης απασχόλησης, τι γίνεται, πληρώνονται λιγότερο και πρέπει να κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, σε λιγότερες ώρες. Αυτό δείχνουν οι στατιστικές Όσο πιο πολύ δουλεύεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά του μισθού. Και αυτό σημαίνει μερική απασχόληση για τις γυναίκες. Αυτό δεν ισχύει βέβαια σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά η κατάσταση είναι πραγματικά ανησυχητική σε πολλά κράτη-μέλη. Δεν θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε ιδιαίτερα για τη μερική απασχόληση. Εμείς αναφερόμαστε κυρίως σε σύγχρονους τρόπους απασχόλησης. Και πραγματικά επαναλαμβάνω εδώ ότι η τεχνική νομοσύνη είναι εξαιρετικά μεγάλη ευκαιρία και δεν πρέπει να τη χάσουμε εμείς οι γυναίκες. Βλέπω την Πρόεδρο να αρχίσει λίγο να αδειμονεί. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ολοκλήρωσα εδώ την ομιλία μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε, για τη συνεργασία. Απαντήσατε στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών πολύ καλά, πιστεύω. Αλλά έχουμε ένα και άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Λυπούμε που δεν έχουμε και άλλο χρόνο. Ελπίζω λοιπόν ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτική ζωή για του γονεί και του φροντιστέ. Έχουμε ένα σχέδιο γνωμοδότηση και θα δώσω το λόγο στην ε, συντάκτρια, κυρία Κουσλόφσκα. E, e, Σα ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω με τον εξή τρόπο. Η πρόταση αυτού του πακέτου περί ισορροπίας ε, μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτικής ζωής είναι ε, μια, ένα διαφορετικό έγγραφο που αντικαθιστά την παλιά οδηγία του 2010 για τις ε, γονικές άδειες. Η αρμόδια επί της επιτροπή είναι η Επιτροπή απασχόληση. Εμείς συντάσσουμε απλώ γνωμοδότηση. Σε αυτή τη χρονοδότηση κατά τη γνώμη μου, η πρόταση της Επιτροπής ε, περιλαμβάνει δύο σημαντικούς πυλώνες ε, που καταρχάς αφορούν την αύξηση της ισορροπίας ανάμεσα στις γυναίκες και στους άνδρες στην αγορά εργασίας. Όσο λοιπόν αφορά αυτούς τους δύο πυλώνες, και κυρίως η ανεπαρξία η η της δυνατότητας μεταφοράς ε, της γονικής άδειας και δεύτερον ε, η δυνατότητα των ανδρών να χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα. Όλα αυτά θα πρέπει λοιπόν να αναδοθούν ως μια ε, επένδυση μακροχρόνια που θα βοηθήσει τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και θα συμβάλλει στην ανεξαρτησία τους. Κατά τη γνώμη μου όμως αυτό θα επιφέρει και οικονομικά ωφέλη γιατί θα υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας. Επίσης θα ήθελα να επισήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η πρόταση αυτή και εμείς έχουμε συμπεριλάβει αυτό το σημείο στη γνωμοδότηση, μιλά για τα δικαιώματα των πατεράδων και για τα καθήκοντά τους εντός της οικογένειας. Θα έπρεπε λοιπόν ε, και μάλιστα ε, εισάγει την ιδέα της γονικής άδειας που είναι υποχρεωτική, θα είναι υποχρεωτική miesiące dla matki, Τέσσερις, μέρες, ε, τέσσερις μήνες για τη μητέρα και τέσσερις μήνες για τον πατέρα χωρίς τη δυνατότητα να μεταφέρονται αυτά τα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει πως περισσότεροι άνδρες θα μπορούν να ε, ε, εκμεταλλευτούν αυτή την οδηγία. Το βασικό πρόβλημα και στις τροπολογίες βεβαίω που καλώ όλους τους συναδέλφους να υποβάλλουν τροπολογίες αν το θέλουν. Δεν θα ήθελα ωστόσο αυτή η γνωμοδότηση να γίνει ιδιαίτερα μακροσκελής. Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε εκείνο το δράμα που υποστήκαμε όσον αφορά την οδηγία για τις ε, άδειες μητρότητας, διότι στο πλαίσιο του Συμβουλίου επικρατούν διάφορες απόψεις για το θέμα τούτο. Ωστόσο θέλουμε η πρόταση αυτή του Κοινοβουλίου να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Άρα λοιπόν, όχι μόνο αυτές, αυτοί οι δύο πυλώνες, η μη δυνατότητα μεταφοράς της γονικής άδεια, αλλά και η μία κατάλληλη αποζημίωση στο ίδιο επίπεδο με την αποζημίωση ασθένειας, αλλά θα πρέπει να δούμε και ε, τι ε, συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που οι περισσότερες απασχολούν ε, πολυάριθμες γυναίκες. Θέλουμε λοιπόν να προστατεύσουμε αυτό το είδος της Ε, στη γνωμοδότησή μου δεν προτείνω κανενός είδους ειδικέ διατάξεις για αυτό το είδος της επιχειρήσης. Μάλιστα θα ήθελα να εξαιρεθούν από, την, από το πεδίο εφαρμογή αυτής της οδηγία. Ωστόσο ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν και αυτό το είδος της εταιρείας στα κάτι μέλη. Νομίζω πως αυτά είναι τα πιο σημαντικά σημεία και θα ήθελα, όπως είπα, να καλέσω όλους τους συναδέλφους να υποβάλουν τις τροπολογίες τους για αυτή την, τροπολογία, για αυτή την ε, οδηγία, συγγνώμη, και να σας καλέσω να στηρίξετε την πρόταση και τη γραμμή που έχω υποβάλει. Στόχος μας είναι η ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες, καλύτερη λειτουργία και συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η άρση των ε, εμποδίων που υπάρχουν στην αγορά για την εργασία των γυναικών, αλλά και να δώσουμε τη δυνατότητα στους πατεράδες, στους άνδρες να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Ακόμα και όσον αφορά την άδεια στους ε, φροντιστές, η πρόταση της ε, Κομισιόν κατά τη γνώμη μου είναι η σωστή και δεν θέλω να υποβάλω ε, τροπολογίες. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα θα δώσω το λόγο στις σκιώδεις, ε, στους σκιώδεις συγκεκριτές. Εγώ ίδια είμαι σκιώδης για αυτό το θέμα. Καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Κοσλόφσκα για το σχέδιο γνωμοδότησής της. Είναι μια πολύ καλή βάση για την περαιτέρω δουλειά μας γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως είπε η Επίτροπος Γιούροβα στη διάρκεια αυτής της θητείας να ληφθεί η οριστική απάντηση για την ισορροπία μεταξύ ε, ιδιωτικής ζωής και ε, επαγγελματικής ζωής. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η εργασία μας και θα πρέπει να συμφωνήσουμε όσον αφορά την, ε, ε, την, την ανυπαρξία δυνατότητας μεταφοράς της άδειας αυτής. Είναι πολύ σημαντικό η μητέρα και ο πατέρας να μπορούν να συμμετέχουν από κοινού σε αυτή τη διαδικασία και αν καταφέρουμε να φτάσουμε σε συμφωνία σε αυτό θα είναι πολύ θετικό. Να επιστήσω ότι την προσοχή σας σε μια άλλη περίπτωση. Υπάρχουν ε, οικογένειες που de facto είναι γονεϊκές, όπου μόνο ένας γονιός ασχολείται με το παιδί, που δεν είναι δηλαδή χωρισμένοι γονείς ή, χωρι... ή σε διάσταση. Γιατί ε, ο... Ε, de facto, εκεί υπάρχει ένας γονιός μόνο που ασχολείται με το παιδί και εκεί πρέπει να προβλέψουμε εξαιρέσεις για αυτές τις περιπτώσεις. Έπειτα, αμοιβή, θα πρέπει να συμφωνήσουμε για μια κοινή θέση σε αυτό το θέμα Η Επιτροπή μας θα οφείλει να απαιτήσει να μείβεται κάθε είδους ε, άδεια με αμοιβή αντίστοιχη της ε, άδεια λόγω ασθενείας. Όμως θα πρέπει να βρούμε μια συμβιβαστική λύση εδώ, γιατί όσον αφορά την, τις αναρωτικές ε, ε, ορισμένοι προβλέπουν το 25% ενώ άλλοι το 100%. Οπότε κάπου πρέπει να βρούμε συμφωνία. Για παράδειγμα 75% ή 85% του μισθού. Ε, έπειτα η προειδοποίηση πριν κάποιος να πάρει την άδεια πατρότητας ή ή μητρότητας. Ε, Πάντω πρέπει να σκεφτούμε κάθε είδου πιθανότητα, γιατί υπάρχουν ας πούμε ασθένειε που δεν μπορούμε εκ των προτέρων να τι προβλέψουμε. Είναι περιπτώσει ανωτέρα βία. Και μπορεί και ποιο να μην μπορεί να ειδοποιήσει εκ των προτέρων. Έπειτα, απαιτήσει αρχαιότητα ή περίοδου εργασία για να μπορεί κανεί να ε, έχει αυτή το είδο την άδεια. Η οδηγία προβλέπει μία τήσια περίοδο. Ε, δηλαδή πρέπει κανεί να έχει εργαστεί για ένα χρόνο σε κάποια εταιρεία για να έχει δικαίωμα άδεια τέτοιου τύπου και δεν ε, γίνεται σαφές αν αυτή η περίοδος μπορεί να θεωρηθεί σωρευτικά, δηλαδή αν κάποιος έχει εργαστεί για ένα χρόνο αλλά σε πολλές διαφορετικές εταιρείες κανονικά θα πρέπει να είναι δυνατόν να ε, προστίθενται αυτές οι χρονικοί περίοδοι εργασίας. Προσοχή τώρα για τις εταιρείε και τις πολύ μικρές εταιρείε ε, εκτός από τις μικρομεσαίες. Καταλαβαίνω πως ε, εκεί η οργάνωση είναι πιο δύσκολη σε περίπτωση που κάποιος ζητήσει τέτοιου είδους άδεια, αλλά απ' την άλλη ε, οι μικρές αυτές επιχειρήσεις τα καταφέρνουν, δεν, μπορούν, δεν, δεν έχουν πολλά προβλήματα γιατί να οργανωθούν καλύτερα. Τώρα, το δικαίωμα που προβλέπεται για τον εργοδότη ε, όσον αφορά τη δυνατότητα να καθυστερήσει τη γονική άδεια. Ε, θα πρέπει η ευθύνη του εργοδότη να είναι περιορισμένη, γιατί δεν μπορεί κανείς να εξαρτάται μόνο από την καλή του θέληση. Και εδώ θα πρέπει να βρούμε κάποια κοινή θέση. Αυτά είχα να πω. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους σκιώδεις. Η ε, κυρία Μπεσέρα πρώτα. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κοσλόφσκα για την εργασία τους που έκανε εδελεχή δουλειά και που ακολουθεί πολύ καλό προσανατολισμό. Το, το σημαντικό είναι τα οι τεχνικές προδιαγραφές να είναι θετικές. Μπορεί να είναι πολύ τεχνικό, αλλά εγώ θα ήθελα να εκφράσω έναν προβληματισμό για το τι οδηγία θέλουμε, ε, τι στόχο έχουμε και από πού ερχόμαστε σε σχέση δηλαδή με, την, με την κατάσταση της γυναίκας. Ποιο είναι ακριβώ ο, ο βασικό στόχο. Το λέει λοιπόν αυτή η έκθεση, το λέει αυτή η οδηγία, διευκόλυνση τη πρόσβαση στην αγορά για τις γυναίκες. Και άρα ξεκινάμε από κάτι που είναι πολιτική επιλογή και φιλοσοφική επιλογή και προγραμματισμός. Πώς δηλαδή θα προσεγγίσουμε από αυτό εδώ το κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους πολίτες, πώς θα προχωρήσουμε με ένα νομοθετικό κείμενο εφόσον δεν μιλάμε για την οδηγία για τη μητρότητα. Μια οδηγία που ισχύει από το 1992, που είναι τελείως ξεπερασμένη και η Κομισιόν μας λέει μόνο ότι το θέμα δεν είναι να προτείνουμε άλλη ή να την αλλάξουμε αλλά να την εφαρμόσουμε 25 χρόνια μετά. Αυτή η οδηγία ε, ισχύει ε, πριν από τη γέννηση του, του γιού μου που είναι 25 ετών. Ε, είναι στα συρτάρια μια οδηγία λοιπόν εδώ και πολύ, πολλά χρόνια και το Κοινοβούλιο πέτυχε τη δέσμευση της Κομισιόν να υποβάλει πρόταση προσαρμοσμένη στην ευρωπαϊκή, σημερινή ευρωπαϊκή κοινωνία. Εδώ δεν έχουμε λοιπόν μια συνολική πρόταση και η Κομισιόν μας λέει ότι δεν λείπει τίποτα, ότι όλα είναι εντάξει. Και έχω την απάντησή σας που λέει ότι αυτό που δείχνει η αξιολόγηση αντικτύπου είναι ότι δεν χρειάζεται επιπλέον νομοθεσία, αλλά χρειάζεται να εφαρμοστεί αυτή που ήδη υπάρχει. Άρα λοιπόν, αν ο δικαιός μας στόχο είναι η ευκαιρία που έχουμε αυτή, αυτό το χρόνο το τόσο κρίσιμο, όπου όλα τα κινήματα σε σχέση με την ισότητα αρχίζουν να συγκλίνουν και έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε μια ε, μεταρρύθμιση προσαρμοσμένη στην κοινωνία, ασχολούμαστε με ένα κομματάκι νομοθεσία για, για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, δηλαδή άδεια αγωνική του μητέρα ή του άντρα στη, μέχρι τα 12 έτη του, του παιδιού ή αν θα δώσουμε μια άδεια στον ε, βοηθό φροντιστή. Όλα πρέπει, εγώ πιστεύω πως θα πρέπει να μιλάμε ε, ε, πιο αποφασιστικά Ξεκολουθούμε να μιλάμε για διαμητρότητες, λες και είναι αναρωτική άδεια, λες και είναι αρρώστια. Ναι, εντάξει, πρέπει να ανακτήσει η γυναίκα. Εδώ μιλάμε όμως και για τα όσα έρχονται μετά. Μέχρι πού να φτάσουμε λοιπόν σε μια σύγκληση ε, για το όταν μιλάμε σε αυτό το κοινοβούλιο τη δυνατότητα να αναθεωρηθεί η οδηγία για την μητρότητα, η αγορά εργασίας ε, θα ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να δέχεται ότι οι γυναίκες δεν είναι πρόβλημα επειδή μπορεί να πάρουν άδεια μητρότητας. Δεν είναι αναρωτική δεν είναι αρρώστια ούτε όταν, κατε, όταν ούτε όταν η μητέρα σου, η οικογένειά σου αποτελείται από δύο πατεράδες, δύο μητέ, μητέρες ή ό,τι θέλεις. Εν πάση περιπτώσει είναι μια άδεια που θα πρέπει να αμείβεται και για πόσο χρόνο και υποχρεωτικά. Εγώ νομίζω πως είναι πολύ θλιβερή αυτή ε, το να μην εκμεταλλευτούμε αυτήν εδώ την ευκαιρία να μιλήσουμε για το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, να διευκολύνουμε τις γυναίκες να μπουν στον κόσμο εργασίας, στην αγορά εργασίας, στις επιχειρήσεις ε, να μπορούν να προσλαμβάνουν γυναίκες και τη δυνατότητα στους πατεράδες να μοιραστούν ε, την γονική άδεια άλλο μητρότητα, άλλο γονική άδεια. Δεν ξέρω, στα αγγλικά μπορεί να σημαίνει άλλα πράγματα, αλλά για, μένα, ε, για τα ισπανικά είναι άλλο πράγμα. Τουλάχιστον ας τοποθετηθούμε πολιτικά σε σχέση με το τι χρειαζόμαστε και για το τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για συνυπευθυνότητα και για ε, μετατροπή της αγοράς και της κοινωνίας για να ε, προσαρμοστεί στον καιρό μας και στην ισότητα και για να καλυφθεί, να γεφυρωθεί το μεσολογικό χάσμα. Ε, τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Βεβαίω, και θα υποβάλλω τι τροπολογίες μου στην κυρία Γκοσλόφσκα σε σχέση με αυτή εδώ τη γνωμοδότηση. πάντω από πολιτική άποψη, πιστεύω πως εδώ σε αυτή την Επιτροπή θα πρέπει να σχηματίσουμε κοινό μέτωπο ώστε να δούμε τι πολιτική ατζέντα θα θεσπίσουμε εδώ περισσότερο αποτελεσματική. Σα ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ορτασούν. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ισπανικά. Πιστεύω πως η πρόταση της Κομισιόν είναι λιγοστή. Εμείς θα θέλαμε να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο. Υπάρχει πρόβλημα και για την κατάθεση τροπολογιών. Γιατί δεν δουλεύουμε πάνω στην οδηγία για την άδεια μητρότητα. Εκεί θα ήταν πιο σφαιρική η προσέγγιση και είναι δύσκολο να προχωρήσουμε εφόσον δουλεύουμε μόνο σε ένα κομμάτι. Έχουμε διάφορες επιλογές, να δούμε τι είναι πιθανό, να, δούμε, να προχωρήσουμε στις ευρωεκλογέ, ξέροντας ποιες είναι οι θέσεις στα κράτη-μέλη. Ε, εάν ζητήσουμε υπερβολικά πράγματα, πιθανότατα θα, δεν, θα πάρουμε, δεν θα πετύχουμε τίποτα να ξεκινήσει πάντως ε, η προσπάθεια απέναντι στο Συμβούλιο για να προσπαθήσουμε κάτι να πετύχουμε. Είναι η, πρώτη, η πρώτη ιδέα οδηγία ε, έμεινε μπλοκαρισμένη και αυτό είναι πολύ κακή αρχή για τον κοινωνικό πυλώνα. Ε, της Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει, αν καταφέρουμε τουλάχιστον αυτό να προχωρήσουμε, θα είναι ένα πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν το θέμα είναι σε επίπεδο Κομισιόν πόσο φιλόδοξοι θέλουμε να είμαστε. Λαμβάνοντα υπόψη ότι η συζήτηση στο Συμβούλιο, αν είναι τέσσερι μήνε, τρει μήνε, σε κάποιε χώρε θέλουν να το κάνουν δύο μήνε, η, πληρωμή, η αμοιβή ε, σε ορισμένα κράτη ε, δεν ε, θέλουν να ακολουθήσουν την πρόταση της Κομισιόν. Οπότε στο Συμβούλιο θα υπάρξουν πολλές πολλές δυσκολίες. Ωστόσο, θα πρέπει εμείς να έχουμε μια ισχυρή θέση ως Κοινοβούλιο στις πιθανές ε, διαβουλεύσεις, έτσι ώστε τουλάχιστον η πρόταση της Κομισιόν να μην αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο και κάποιες προτάσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ένας από τους κύριους στόχους της πρότασης είναι περισσότεροι άνδρες να αναλάβουν την ευθύνη τους απέναντι στο παιδί τους. Αυτός είναι ένας κύριος ε, στόχος. Δεν είναι άδεια πατρότητας λοιπόν, η οποία θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική. Αυτό το μήνυμα θα πρέπει να βγει από το, το κοινοβούλιο, ότι δηλαδή εφόσον πρόκειται για μια αγωνική άδεια που είναι περιορισμένη χρονικά, ε, να είναι τουλάχιστον υποχρεωτική. Και η αποζημίωση για αυτές τις μέρες να είναι στο επίπεδο που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να είναι αντίστοιχη τουλάχιστον με την αμοιβή στη διάρκεια της αναρωτικής άδειας. Ε, και τα κράτη-μέλη δεν θα το επιθυμούν αυτό, ε, γιατί αυτές καθορίζουν. Ας πούμε, στην Ισπανία έχουμε 80% της αμοιβή ε, και είναι αρκετά ψηλό. Εγώ πιστεύω πως θα πρέπει ωστόσο να το θεσπίσουμε, ώστε να υπάρχει μια πλήρης αμοιβή στην περίπτωση που κανείς πάρει αυτή την άδεια. Γιατί διαφορετικά, όσο πιο ψηλό επίπεδο αμοιβή, τόσο περισσότεροι άντρε θα πάρουν αυτή, θα ζητήσουν αυτή την άδεια. Το πρόβλημα ε, που θα έχουμε αν το, αν, δεχτούμε εδώ ε, είναι ότι στην οδηγία για την άδεια μητρότητας ε, η αμοιβή είναι η ίδια με τη, αυτή της αναρωτικής άδεια. Γι' αυτό και είναι προβληματικό το να ασχολούμαστε με ένα κομμάτι μόνο αυτού του τύπου άδεια. Ανάλογα λοιπόν με το πώς θα καταλήξει αυτή η οδηγία μετά τους ε, τριμερείς ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε μια μεταρρύθμιση της άδεια Μητρόπιτας, γιατί μπορεί να βρεθούμε σε ε, κατάσταση αβεβαιότητας. Λοιπόν κλείνω γιατί αρχίζω και μακρηγορώ. Πάντως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να περάσει. Ξέρουμε ότι στο Συμβούλιο είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά ως Κοινοβούλιο πρέπει να πάμε με μια φιλόδοξη πρόταση, πιο φιλόδοξη από τις Κομισιόν. Και στα στοιχεία που ανέφερα νομίζω πως υπάρχουν δυνατότητες ώστε αυτό το πακέτο να είναι πολύ φιλόδοξο. Κύριε Κουνέμα. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Ανέτσικα Κοσλόφσκα για την δουλειά που έχει κάνει. Πριν προχωρήσω στο σχόλιο μου επί των τροπολογίων, θα πω ότι συμφωνώ με όσα είπε η συνάδελφος Μπερέσα για το πολιτικό διακύβευμα, Μπεσέρα. Έχω και εγώ στο παρελθόν τοποθετηθεί ανάλογα και δεν γίνεται κάθε φορά να θέλουμε να ανοίξει το θέμα αυτό, όταν θέλουμε να ανοίξει το θέμα αυτό, να μας κουνάνε το δάχτυλο κάποιοι συνάδελφοι και να μας λένε πώς ονερβαθούμε. Αλλά και να μας λένε να μην στοχεύουμε ψηλά για την πρόταση αυτής της οδηγίας. Δεν νομίζω ότι το Κοινοβούλιο είναι εδώ για να εκφράζει θέσεις αρεστές στο Συμβούλιο. Είμαστε εδώ για να εκφράζουμε τους πολίτες της Ευρώπης. Και οι πολίτες θέλουν αλλαγές εμείς ως ομάδα της αριστεράς θα προτείνουμε τις απαραίτητες αλλαγές χωρίς φόβο και με πολύ πάθος. Ε, πολλές από τις τροπολογίες της ε, εισηγήτριας με βρίσκουν σύμφωνοι ως προς το πνεύμα και την κοινική τους κατεύθυνση. Για παράδειγμα, η τροπολογία 1, στην οποία μιλάει η εισηγήτρια την ανάγκη ποιοτικών δομών φροντίδας για τα παιδιά και τα εξαρτημένα μέλη της οικογένειας. Η τροπολογία 13, στην οποία η συγκήτρια σωστά λέει πως το δικαίωμα της άδειας πατρότητας πρέπει να επεκταθεί και για τους πατεράδες οικογενειών που υιοθετούν παιδιά. Συμφωνώ επίσης και με την τροπολογία 27 που εισάγει ρήτρα μη υπαναχώρησης δίνοντας έτσι έμφαση στο ότι οι διατάξεις της οδηγίας θέτουν το ελάχιστο, το μίνιμουμ που θα πρέπει να υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τυχόν ενισχυμένα δικαιώματα που ισχύουν τώρα και σε κάποια κράτη-μέλη δεν τα υποχωρήσουν. Στις τροπολογίες της κίτριας υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία με έβαλαν σε σκέψη είμαι ανησυχήσαν. Προσωπικά λέω ναι στις καλύτερες και ποιοτικέ υπηρεσίες φροντίδας, αλλά όχι όταν αυτό χρησιμοποιείται για να γίνει ακόμα πιο ελάχιστο το ωράριο εργασίας των γονέων. Δεν λέω ότι έτσι σκέφτηκε η συγγήτρια. Έχω ακούσει όμως τις θέσεις των εργοδοτών και της ε, Business Europe και εκείνοι είμαι σίγουρη ότι έτσι θα το ερμηνεύσουν. Γιατί αυτό υπονοούσαν πίσω από τις θέσεις που μας κοινοποίησαν. Ένας γονιός που θα πρέπει να αφήσει το παιδί του σε μια μονάδα φροντίδας η οποία θα λειτουργεί πέραν του λογικού ωραρίου φυσικά δεν θα μπορεί να αρνηθεί στον εργοδότη του να μείνει μία και δύο ώρες παραπάνω στη δουλειά. Επί αυτήν την έννοια μπορεί να ελαστικοποιήσει ακόμα περισσότερο το ωράριο των εργαζομένων και αυτή τη φορά όχι προ όφελο τη προσωπική αλλά και τη επαγγελματική ζωή του. Άλλε τροπολογίε που με έβαλαν σε σκέψη είναι τροπολογία 2 που λέει πω θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο δια, διάστημα εργασία ενό έτου πριν ο εργαζόμενο μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματο τη γονική άδεια και η τροπολογία 3, όπου η συγκήτρια αναφέρει πω θα πρέπει να υπάρχει μια εύλογη χρονική περίοδο προειδοποίηση από τον εργαζόμενο στον εργοδότη ότι θα κάνει χρήση του δικαιώματο του η γονική άδεια. Μπορεί να μα πει η συγκήτρια πώ η ίδια αντιλαμβάνεται το εύλογο διάστημα, άραγε Μπορείτε να μας πείτε γιατί θέλετε να περιορίσετε το δικαίωμα για γονική άδεια μόνο σε εργαζόμενους που βρίσκονται σε υπηρεσίες για τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο μάλιστα ορίζεται το μέγιστο σε ένα έτος. Αρκετά έχουν απορριθμιστεί οι σχέσεις εργασίας. Μην συμβάλλουμε στο να δημιουργηθούν εργαζόμενοι δύο και τριών ταχυτήτων. Επίσης, η τροπολογία 24 έχει μια καλή ιδέα ως βάση, αλλά οι λέξεις με τις οποίες περιγράφεται, η ιδέα αυτή δεν με βρίσκουν σύμφωνη. Πιστεύω πως αποδυναμώνεται η κατοριστική και ουσιαστική συμβολή που μπορούν να έχουν οι συλλογικέ συμβάσει για την επίτευξη των σκοπών τη οδηγία και για την ομοιογενή εφαρμογή τη. Ναι, μπορούν να συμβάλλουν στην εξισορρόπηση προσωπικής επαγγελματική ζωής και να μπορούν να προάγουν και να διασφαλίζουν την ισότητα στον χώρο εργασία και το λέω έχοντα εμπειρία από τη χώρα οικογική μου στην Ελλάδα. Τέλο, θα... για να αφήσω χρόνο και στου υπόλοιπου συνάδελφου, δεν θα σχολιάσω λεπτομέρειε τη υπόλοιπε τροπολογίε. Έτσι κι αλλιώ έχουμε διαφορετικέ απόψει για το θέμα του προσωπικού προσαρμόσιμο χρόνο εργασία το επίπεδο αμοιβή των γονικών αδειών, της ηλικία των παιδιών, των φροντιστών. Ελπίζω να καταφέρουμε να βρούμε μια κοινή λύση και να καταλήξουμε σε μια δυνατή διαπραγματευτική εντολή για το νομοθέτημα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σουσίνκη. Μόνο για δύο λεπτά παρακαλώ, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Έχουμε ακόμα ένα ζήτημα πριν από τη συνάντηση των συντονιστών. Λυπάμαι. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μην ανησυχείτε, δεν θα με Πράγματι συνεργάστηκα ε, με την συγγήτρια για αυτή την ε, γνωμοδότηση και την ε, ευχαριστώ γιατί υιοθέτησε και έλαβε υπόψη πολλές από τις ε, προτάσεις μας, ιδίως για τις πολύ μικρές και μικροψές επιχειρήσεις που με την οδηγία αυτή θα χρειαστούν πολύ περισσότερη ευελιξία και χωρίς να μιλάμε και για το κόστος που εμπλέκεται εδώ. Υπάρχει μια διαφορά με την εισηγήτρια, από ό,τι φαίνεται και με άλλους, σε ό,τι αφορά την φορητότητα του δικαιώματος της γονικής άδειας και δυνατόν μεταβίβαστες δηλαδή ε, σε άλλον, να τους έχουν το δικαίωμα να κάνουν, να πάρουν αυτή την άδεια, ε, πράγματι μπορούν να το ασκήσουν, όμως ε, με το να τους λέμε ότι δεν μπορούν να τη μεταβιβάσουν, γίνεται αυτό το δικαίωμα υποχρέωση. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι μια απόφαση του ζευγαριού και εσείς de facto την ε, καθιστάτε υποχρεωτική σαν διάταξη, γιατί στην οδηγία προβλέπεται ένα διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών. Το διάστημα κάτω των τεσσάρων μηνών δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, οπότε θα είναι όχι τόσο δικαίωμα όσο υποχρέωση. Και δεν συμφωνώ σε αυτό. Φυσικά θα συνεργαστώ με όλους προκειμένου να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω ένα μόνο σημείο. Η Επίτροπος πριν από λίγο εδώ μας μίλησε για την οδηγία, την προηγούμενη οδηγία, η οποία δεν πέρασε στο Συμβούλιο και θα αντικαταστήσει αυτό το οποίο ουσιαστικά συζητάμε σήμερα την ε, οδηγία αυτή. Τελικά λοιπόν αυτό που βλέπουμε ότι όσον αφορά την ε, στήριξη και τα συνοδευτικά μέτρα για τις έγκυες γυναίκες και τις ε, διακρίσεις που συνεχίζουν να γίνονται. Όπως είπε η κυρία Μπέσερα, πρέπει να μιλήσουμε λίγο και για θέματα υγείας των γυναικών. Η γυναίκα μετά τον τοκετό χρειάζεται λίγο χρόνο να ανακτήσει την προηγούμενη κατάσταση και βεβαίως είναι πολύ σημαντικά τα θέματα της ε, άδειας αυτής. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για υποχρέωση να πάρει κάποιος μια τέτοια άδεια, αλλά πρέπει να δούμε ειδικότερα τα θέματα υγείας και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και μετά τον ε, το κετό. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρωθούμε σε αυτά και να δούμε πώς ακριβώς θα τα ενσωματώσουμε σε αυτή την οδηγία. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή. Υπάρχει κάποιος εδώ από την Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Να σας πω ότι η Επιτροπή είναι πολύ ευτυχής με το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής, το οποίο θεωρούμε πάρα πολύ εμπεριστατωμένο και αντικατοπτρίζει τα κύρια σημεία της πρότασης της Επιτροπής και το πνεύμα εμείς βεβαίως και συμφωνούμε με όλα αυτά που ακούσαμε. Το θέμα παραδείγματο χάρη είναι το πώς θα υλοποιηθεί αυτή η πρόταση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μην υπάρχει τεράστιος αντίκτυπος. Καταλαβαίνουμε αυτό που λέει η συγγήτρια, Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Βεβαίως ε, έχω και κάποια άλλα τεχνικά σχόλια, αλλά θα τα συζητήσουμε κατευθείαν με την εισηγήτρια, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Κόσλοφ Πολύ, πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους που πήραν το λόγο. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας και φυσικά και θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Ακούσαμε ότι υπάρχει βούληση για σύγκληση, για κοινή εργασία. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε κοινέ προτάσεις εκεί που γίνεται, να πλησιάσουμε δηλαδή τις διαφορετικές μας προσεγγίσεις όταν αυτές είναι διαφορετικές. Η κυρία Ζαμπόρσκα είπατε ότι αμφισβητείται το θέμα της πιθανής, αν θέλετε, αντικατάστασης της οδηγίας που αφορά την προστασία των μητέρων από αυτή την οδηγία. Δεν έχει καμία σχέση. Βέβαια τα θέματα είναι συναφή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται αυτή εδώ η οδηγία να αντικαταστήσει την άλλη. Εδώ μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Μιλάμε για τους ε, γονείς και θέλουμε να ξαναδούμε τους κανόνες ε, που ισχύουν. Καμία σχέση, επαναλαμβάνω, με την οδηγία την οποία δεν την ακουμπάμε που αφορά την προστασία των μητέρων. Αυτή η οδηγία που αφορά τον χρόνο και τις άδειες των γονέων, αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Άλλο κείμενο και άλλη νομική βάση, αλλά άλλο σκεπτικό αν θέλετε. Πιστεύω ότι όπως και άλλοι εξάλλου που πήραν το λόγο, θα πρέπει με αυτήν την πρόταση που κάνουμε σήμερα να πετύχουμε κάτι και στη συζήτησή μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με το Συμβούλιο. Γι' αυτό και λέω ότι αυτό το κείμενο το οποίο περιέργως το συζητάμε πριν από την οδηγία για την προστασία των ε, μητέρων είναι κάτι το οποίο το περιμένουν οι πολίτες από μας. Σε γενικές γραμμές η οδηγία αυτή θα θέσει τα κατώτερα όρια. Αυτό δηλαδή θα πρέπει κατελάχιστον να ισχύει στα κράτη-μέλη. Και αν παραδείγματο χάνει σε μια χώρα υπάρχει μεγαλύτερη, αν θέλετε, πρόβλεψη για τη διάρκεια της γονικής άδειας, δηλαδή τέσσερις μήνες και τέσσερις μήνες οκτώ μήνες, θα πρέπει αυτό να μπορεί να παραμείνει. Είμαστε ευέλικτοι, αλλά θέτουμε απλώς τα ελάχιστα τα οποία θα πρέπει να ισχύουν. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα ε, γονικής άδειας. Για τις χώρες αυτές που έχουν είτε μικρότερη διάρκεια είτε καθόλου. Και βεβαίως και ε, προσφέρουμε μια δυνατότητα να πάρουν οι γονείς γονική άδεια. Δεν είναι υποχρέωση. Τους δίνουμε το δικαίωμα να το κάνουν και σε καμία περίπτωση δεν τους υποχρεώνουμε. Ούτε τη μητέρα ούτε τον πατέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες σας τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Να πω μόνο ότι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι 10 Απριλίου στις 5 το απόγευμα. Θα εξετάσουμε ε, τις 14 14-15 Μαΐου και θα ψηφιστεί στην ε, Επιτροπή 28 Μαΐου. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημέρας διάταξης, η κατάσταση στην Ουγγαρία. Έχουμε ένα σχέδιο νομοδότηση τη κυρία ε, Μαρία Νόχιλ. Ο κύριο Μαχτά ε, την αντικαθιστά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπω είπατε, η Μαρία Νόιχλη δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα και μου ζήτησε να σας διαβάσω τις παρατηρήσεις της, με τα χαράς να το κάνω. Γι' αυτό και θα μιλήσω σε πρώτο πρόσωπο, ακόμα και αν αναφέρεται σε γυναίκα. Ως ε, εισηγήτρια ε, της Επιτροπής για την ε, τρέχουσα κατάσταση στην Ουγγαρία, είχα την τιμή πριν από μερικές εβδομάδες να πάω στην Ουγγαρία μαζί με άλλα μέλη της Επιτροπής. Παρότι ήταν πολύ έντονη η εργασία μας και το πρόγραμμά μας ήταν φορτωμένο με πολλές συναντήσεις, με ακτιβίστριες, με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, είμαι σίγουρη ότι δεν μας δεν καταφέραμε να ε, έχουμε μια απόλυτα συνολική εικόνα της κατάστασης. Θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω ορισμένα στοιχεία που με προβληματίζουν και θα πρέπει να ενταχθούν στη γνωμοδότηση. Πρώτον, υπάρχει μια ε, υπαναχώρηση και επανερμηνεία ε, της πολιτικής για την ισότητα των φύλων και η η νομοθεσία του 2010 δεν εφαρμόζεται. Ο αντίκτυπος των οργανώσεων που χρηματοδοτούνται από ξένες χώρες, αλλά και ευρωπαϊκές, ε, περιορίζουν σημαντικά την ε, εμπλοκή της κοινωνία των πολιτών και τη λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η υπονόμευση της, ε, των πολιτικών και άλλων ελευθεριών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερως. Τρίτον, ε, η επίθεση κατά των δικαιωμάτων της ε, αυτοδιάθεσης των γυναικών στην απαραγωγική τους υγεία είναι ξεκάθαρη. Η πρόσβαση στην ε, έκτρωση είναι όλο και πιο δύσκολη. Επίσης, δυσκολίες υπάρχουν και για τις αγγείους και υπάρχει σημαντική δίευση και διάκριση των Ρωμά σε συγκεκριμένου τομεί. Είναι ένα από τα σημεία που θεωρώ πολύ σημαντικά στην νομοδότηση 11 Απριλίου βέβαια είναι η, υποβολή, προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών. Ε, αν και αυτό είναι πολύ σύντομα βέβαια. Σας ευχαριστώ για την συνεργασία. Ευχαριστούμε κύριε Μαχτά. Να δώσουμε τώρα το λόγο ε, στους εσκιώδες, η κυρία Ζαντόφσκα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό παρακαλώ να σας ενημερώσω ότι ε, αυτό το τμήμα της συνάντησής μας ε, καταγράφεται από τα ουγγρικά μέσα ενημέρωσης και θα ήθελα να ρωτήσω τα μέλη εάν ε, έχουν αντίρρηση με αυτή την μαγνητοσκόπηση. Παρακαλώ. E, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως, σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Η δική μου πρόθεση είναι να είμαστε φιλόδοξοι και θα προσπαθήσουμε να υποβάλουμε τροπολογίες απαιτητικέ γιατί δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτά που συμβαίνουν χωρίς να αντιδράσουμε ούτε στην Ουγγαρία ούτε στην Πολωνία. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι η πολιτική για την ίση μεταχείριση δεν είναι κατά της πολιτικής για την οικογένεια. Μπορεί να συμπληρωθούν και σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να ανταποκριθούμε και στις ανάγκες των οικογενειών, δηλαδή των ανδρών και των γυναικών. Έχω την εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την υποχρέωση να δει ακριβώς ποια είναι η χρηματοδότηση των ε, φορέων αυτών και των συλλόγων που κάνουν λόμπι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με ποιο τρόπο κάνουν λόμπι, ποιος τους στηρίζει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουσιαστικά δεν κατονομάζει αυτούς που κάνουν λόμπι εδώ σαν πράκτορες. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε λοιπόν να στηρίξουμε κάποιον ο οποίος ουσιαστικά δεν τηρεί ναι. τις συστάσεις που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμάς δεν είναι αρμοδιότητά μας να παρακολουθήσουμε την υλοποίηση και να επιβάλλουμε κανενός είδους ε, κυρώσεις. Αλλά μπορούμε να αξιολογήσουμε την υλοποίηση, μπορούμε να περιοριστούμε στις αρμοδιότητες ε, της Επιτροπής μας και γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι καθοριστικό να συμπληρωθεί αυτή η έκθεση με κάποιες άλλες προτάσεις για την ίση μεταχείριση και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ, κυρία Βυσνεύσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Ως ε, εισηγήτρια της ε, γνωμοδότησης ε, από πλευράς στερετικών μεταρρυθμιστών να πω ότι δεν στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου για αυτή την έκθεση σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ουγγαρία. Ε, οι Βρυξέλλες δεν συμφωνούν με τον τρόπο που λειτουργούν τα, τα κρατημέλη. Αλλά εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό, δεν συνεργαζόμαστε με τους δικτάτορες των Βρυξελών, δεν έχει καμία αρμοδιότητα ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Βρυξέλλες ευρύτερα να ε, παρεμβαίνουν στα εσωτερικά μας. Μπορούμε μόνο ο καθένας να λειτουργεί με βάση τις ε, αρμοδιότητες που το έχουν εκχωρηθεί. Επιπλέον, τα κράτη-μέλη ε, εφαρμόζουν διαφορετικές κοινωνικές πολιτικές βάσει παραδόσεων και αξιών. Και ακριβώς αυτή η πολυμορφία δεν είναι αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως, εγώ θεωρώ ότι αυτή η πολυμορφία είναι το δυνατό σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η αποτελεσματική λειτουργία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συνάδει με τον σεβασμό προς αυτή την πολυμορφία και προς τις αξίες που είναι, που σημαντικές για τις κοινωνίες των κρατών μελών και δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν οι Βρυξέλλες σε, σε αυτές τις αξίες, όπως για παράδειγμα η οικογενειακή ζωή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να μπαίνει σε ξένα χωράφια σε επίπεδο που δεν είναι απαραίτητο γιατί αυτά πρέπει να τα αφήνουμε στην επικουρικότητα. Κατανοώ πραγματικά ότι αυτό είναι επισήμω και τυπικώ μία διεύρυνση των ερμοδιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθεί λοιπόν μέσω αυτή τη νομοδότηση η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί με ζητήματα ε, που δεν ε, έχει λόγο να ασχοληθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκεται στα εστερικά της ε, Ουγγαρίας, επικρίνει τις αξίες ε, της ουγγρικής κοινωνίας και αυτό ε, δεν είναι σωστό. Όπως προκύπτει και από τα στατιστικά στοιχεία, βλέπουμε ότι η κατάσταση των γυναικών στην Ουγγαρία δεν εμπνέει μεγαλύτερη ανησυχία από τις άλλες χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά υπάρχουν και ζητήματα στα οποία θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο η Ουγγρική κυβέρνηση, όπω η συμμετοχή των γυναικών ε, ε, στι θέσει ευθύνη στην αγορά εργασία, καθώ ε, και η συμμετοχή τους σε υψηλές κυβερνητικές θέσεις, αλλά και άλλα προβλήματα όπως το μισθολογικό χάσμα, η βία κατά των γυναικών, Εκεί είναι απόλυτο συγκρίσιμα τα στοιχεία με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να μείνει λοιπόν έξω από τα εσωτερικά μας ζητήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά, στην οδηγία για την εξισορρόπηση προσωπικού και επαγγελματικού βίου, και εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ουγγαρία. Ούτε έχουν ολοκληρωθεί βέβαια οι ε, εργασίες επί της οδηγίας. Πρέπει επίσης να καταλάβετε ότι η Ουγγαρία εφαρμόζει ε, ενεργώς μία πολιτική οικογενειακού βίου που στηρίζει ε, τους ε, άντρες και γυναίκες που επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Οπότε ήδη εφαρμόζει η Ουγγρική κυβέρνηση φιλική προς την οικογένεια νομοθεσία. Είδαμε σημαντική μείωση των αμβλώσεων στην Ουγγαρία τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει σχέση ακριβώς με αυτή την ενεργό ε, και πολύ στοχευμένη οικογενειακή πολιτική στην Ουγγαρία. Υπάρχει ε, πολύ καλή άδεια μετρότητα στην Ουγγαρία και σημαντική στήριξη προς τους νέους και στις νέες οικογένειες για τα στεγαστικά δάνεια και για άλλα ζητήματα. Ε, στη γνωμοδότηση αυτή, όπως και σε κάθε έγγραφο της, της Επιτροπής ΦΕΜ, ε, αναφέρεται η κύρωση της, ε, της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης. Πάντα γίνεται αυτή η παρότρινση, λες, και είναι Ευαγγέλιο αυτή η σύμβαση. Ε, επιπλέον, ε, γίνεται πάλι αναφορά στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κατάχρηση της θέσης μας για να μιλούμε για σεξουαλικές και αναπαραγωγικές ελευθερίες, γιατί αυτές είναι ξεκάθαρα αποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γκαρθία Πέρε. παρακαλώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά δεν ισχυρίζεται ότι είναι ο κύριος των πολιτικών ε, για τον ε, αγώνα κατά της ανισότητας μεταξύ των φύλων. Εμείς υποστηρίζουμε τη σύμβαση της Ισταμπούλ και μάλιστα θεωρούμε πως ο αγώνας αυτός θα πρέπει να γίνεται από όλους και από όλες ε, τα επίπεδα και τα ευρωπαϊκά όργανα και από τις εθνικές κυβερνήσεις επίσης. Γι' αυτό πιστεύω πως είναι κάτι σημαντικό και για να τελειώσω όσον αφορά τα αρμοδιότητες, το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να νομοθετεί η Ευρώπη και να αποφασίζει. Εγώ καταλαβαίνω πως σε αυτή την έννοια υπάρχουν διαφορετικές θέσεις. Ωστόσο, κανείς δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Ε, μπορούμε λέει, να μιλάμε για τις οικογενειακές πολιτικές, αλλά όχι για τις ελευθερίες των γυναικών. Εγώ θεωρώ πως η ελευθερία και η ισότητα είναι θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αξίες ε, και άκουσα μάλιστα, ε, ε, τα σας αναφέραμε εδώ σε αυτές τις παρεμβάσεις. Αν ελευθερία λοιπόν των γυναικών είναι αξία των ευρωπαϊκών θεσμών, άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα θα πρέπει να εγγυηθούν την ελευθερία όλων των γυναικών σε όλες τις χώρες. Και εντό αυτής της ελευθερίας εντάσσεται και η ελευθερία να γίνει καμία μητέρα ή όχι και την ελευθερία να προσέξει τα αντισυλληπτικά μέσα. Δεν μπορεί στον 21ο αιώνα να υπάρχουν χώρες όπου δεν είναι εγγυημένε αυτές οι ελευθερίες. Σας ευχαριστώ. Κύριος Μάρτης. Ευχαριστώ. Μπορώ να μιλήσω. Η Μαρία Νόγελ ανήκε στην αντιπροσωπεία που πήγε στην Ουγγαρία. Εδώ το θέμα μας δεν είναι να πούμε πράγματα υπέρ του Ορμπάν ή όχι. Να πούμε αν αυτά που διαπίστωσε ισχύουν ή όχι. Φαντάζομαι ότι συνάντησε ανθρώπους ε, από την κοινωνία των πολιτών που ζουν εκεί, που πολεμούν για τα δικαιώματα των γυναικών δεν τα έβγαλε από το μυαλό της, αν θέλετε, αυτά που λέγει την Ουγγαρία. Συνάντησε άτομα, προσωπικότητες, μικιό, συλλόγους, ενώσους. Άρα το ερώτημά μας είναι αυτό. Το αν θεωρεί η Ουγγαρία, αν θέλετε, ότι αυτές οι αξίες είναι ε, αξίες για τις οποίες πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ας διαβάσει τις συνθήκες η Ουγγαρία και ας ε, θέσει τα κριτήρια. Κυρία Μπεσέρη, μόνο δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ σύντομα, γιατί πολλοί πήραν το λόγο. Εγώ εκπροσωπώ την κυρία Μολινάρ, που δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Δεν είναι μάλλον σε θέση να συμμετάσχει. Θα ήθελα μόνο να αναφερθώ στα συμπεράσματα της επίσκεψης ε, στη Βουδαπέστη. Ε, πήρε η κυρία Γιουρόχα και η κυρία Νόχελ. Έχουν συνεργαστεί συμπεράσματα μετά από συναντήσεις με ΜΚΟ, με οργανώσεις ε, ε, που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των γυναικών. Αυτές λοιπόν οι οργανώσεις λένε ότι βρίσκονται, ε, δέχονται επίθεση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους. Αυτές πρέπει να ακούσουμε λοιπόν. Εκείνες που λένε ότι υπονομεύονται τα δικαιώματά τους. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε κατά νου τα ευρήματα ε, αυτής της ε, έκθεσης και οι φιλελεύθεροι θα υποβάλουν τροπολογίε με συγκεκριμένα ερωτήματα. Για παράδειγμα, γιατί η Ουγγαρία είναι τόσο χαμηλά σε ό,τι αφορά τον ε, δίκτυ ισότητας των φύλων. Πρέπει λοιπόν να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει και γιατί δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία για την ισότητα των φύλων. Πρέπει να τεθούν αυτά τα ερωτήματα. Γιατί όλο ένα και λιγότερες γυναίκες συμμετέχουν σε θέσεις ευθύνης γιατί υπάρχουν ε, ε, επιθέσεις κατά της ε, έρευνας και κατάρτισης, γιατί υπάρχει περιορισμός της ελευθερίας έκφρασης. Και επίσης να αναφέρω ότι η ευρωπαϊκή κυβέρνηση θέλει να φτιάξει δική της εκδοχή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, αφήνοντας εκτός τη διάσταση του φύλου, που είναι τελικά το, όλο, όλο σκοπός της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης εφόσον προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει και να τη σέβεται, για να σέβεται τις αξίες της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεματοφύλακα αυτών των αξιών. Η Αγγέλικα ανέφερε κάτι ενδιαφέρον εδώ. Πρέπει να συγχαρούμε τον Ανδρέα Πέτερ από το Central European University που έλαβε ε, ένα ευρωπαϊκό βραβείο το 2018 για ε, τις ε, αξίες αυτές. Ε, συναντηθήκαμε με την νικήτρια και είναι πραγματικό σημείο αναφορά. Θα πρέπει να την ακούσουμε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η κυρία Ward. Εγώ δεν ήμουν στην αποστολή, αλλά έχω πάει στην αποστολή με τη Μαρία Νόιχλη στο παρελθόν και ξέρω ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος, συμπονετικός. Είχαμε πάει μαζί στο Μόναχο σε μια αποστολή για να δούμε πώς ε, υποδέχεται η Γερμανία τους πρόσφυγες και πήγαμε και σε μια διεθνή αποστολή στο Μαλάουι, όπου ε, συναντήσαμε τρομερά ευάλωτες ε, γυναίκες ε, που ζουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτιστικό περιβάλλον και κουλτούρα. Οπότε είμαι απολύτως βέβαιη ότι η έκθεση της κυρία Νόιχλ είναι ακριβής και δεν παρεμηνεύει τα όσα είδε. Τώρα σε ό,τι αφορά την παρίσφρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κατά πόσο μπλέκεται στα της Ουγγαρίας. Δεν είναι ότι μπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι θέμα συνεργασίας και ανταλλαγής βέλτιστων των πρακτικών. Αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, καθόμαστε όλοι μαζί στο δύο τραπέζι, ε, συζητάμε μεταξύ μας, μαθαίνουμε ένας από τον άλλον και ουσιαστικά κατανοούμε ότι βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, ότι αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις και στην Ευρώπη και εκτός και ότι αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε επί συγκεκριμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχουν ήδη συμφωνηθεί γιατί εμπεριέχονται στην ε, συνθήκη, ε, δεν γίνεται να διαλέξετε αλλά ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό κάνει το Βασίλειο. Θέλουμε αυτό, θέλουμε εκείνο, το άλλο όμως όχι. Θέλουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά όχι τους κανόνες. δεν γίνεται. Γιατί έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είναι μια ένωση ε, αξιών. Ε, Θέλω να δω τι ακριβώς θέλουν οι νέοι. Και για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων πρέπει ακριβώς να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές τι νέες γυναίκες που ε, βγαίνουν προς τα έξω και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα πραγματικό αγώνα ε, για τις προοδευτικές αξίες στον 21ο αιώνα. Και πραγματικά φοβάμαι ότι εάν δεν λάβουμε υπόψη τη σημασία ε, της, ε, των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, θα χάσουν τη ζωή τους γυναίκες. Γιατί αυτό είδαμε στο Μαλάουι. Δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση. Δεν καταλαβαίνουν ε, τον οικογενειακό προγραμματισμό. Χάνουν τη ζωή τους γυναίκες και παιδιά λοιπόν εξαιτία αυτού και εγώ δεν θέλω να λάβω αυτή την ευθύνη και να τις πάρω στο λαιμό μου. Ευχαριστώ πολύ. Να σα ενημερώσω ότι η προθεσμία κατάθεση των είναι η 10η Απριλίου μέχρι τις 11 το πρωί. Θα ψηφίσουμε στη ΦΑΜ 14-15 Μαΐου. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να πω μόνο ότι η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 12 Απριλίου στις 9 το πρωί. Ευχαριστώ. Σε μερικά λεπτά ξεκινούμε τους, ε, τις συνεδρίες των συντονιστών και το θύρον. <laughs> Okay, okay.